But maybe next time we don't use them in at all. No, well, or to incorporate Benson, Benson yeah, exactly. because it's uh, uh, efficiency of building. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσουμε θερμά τον Επίτροπο Μοέντας, που για μια ακόμη φορά επισκέπτεται την Επιτροπή μας. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε για έναν ακόμη διαρθρωμένο διάλογο μαζί σας για πολύ σημαντικά θέματα. Πρόκειται για τα βασικά πορίσματα μετά από την εσωτερική αξιολόγηση του ορίζοντα 2020. Πολύ σημαντική αυτή η αξιολόγηση και επίσης το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, ένα εξίσου σημαντικό θέμα για μας, ε, και το μελλοντικό πρόγραμμα του 2018. Αυτά μαζί με την αδιάμεση αξιολόγηση του, του ορίζοντα 2020 είναι ζητήματα μείζωνος σημασίας. Επίσης, ε, να επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις υιοθέτησε το ψήφισμά του για τον ορίζοντα 2020 και την έκθεση εφαρμογής που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Οι εκθέσεις εφαρμογής είναι ένα νέο τρόπο να εξακριβώσουμε αν οι νομοθετικέ μα προτάσει λειτουργούν και στι περιφέρειες. Ξεκίνησε με μελέτη, αποστολέ, ακροάσει και περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση όχι μόνο της έμπρακτης εφαρμογής του ορίζοντα 2020 αλλά ατενίζει και το μέλλον και περιέχει σαφείς ιδέες, απόψεις και προτάσεις για το μέλλον κυρίως για το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο υπερθμών 9, δηλαδή για την περίοδο μετά το 2020. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα αυτά για μας κύριε Επίτροπε. Και θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο για να μας εξηγήσετε πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την ενδιάμεση αξιολόγηση και να μας παρουσιάσετε και το μελλοντικό σας σχέδιο εργασιών για το 2018 και 2000, 2020 και το, την πρόταση για το FP9, το ένα το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο που θα υποβληθεί. μετά το 2019. Μας ενδιαφέρουν οι προτάσεις σας για μετά το 2019, γιατί μόλις δύο χρόνια μας χωρίζουν από τις επόμενες ευρωεκλογέ, οπότε θέλουμε να σχηματίσουμε εντύπωση και για το μελλοντικό σας πρόγραμμα και για τις προτάσεις σας για το ένατο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο που θα πάει μέχρι το 2027. Ευχαριστώ. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να συζητώ μαζί σας. Είστε η Επιτροπή μου, έτσι σας αποκαλώ. Ελπίζω ότι δεν σας ενοχλεί, αλλά πάντα είναι χαρά να συζητώ μαζί σας για το μέλλον και να σας ενημερώνω για την εργασία που είναι υπό εξέλιξη, τις εργασίες μας που είναι υπό εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα την προηγούμενη εβδομάδα και σας ευχαριστώ γι' αυτό Είχαμε πολύ επικοδομητικό διάλογο και συζητήσαμε την έκθεση Καμπεθών Ροήθη στο Στρασβούργο και την έκθεση Σακοράφα για το πρίμα και με χαροποίησε ιδιαίτερα στην εργασία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εργασία σας για το πρίμα. Νομίζω ότι η Κομισιόν έκανε το καθήκον της, αλλά κάναμε το καθήκον μας χάρη σε εσά που μας βοηθήσατε για να διαμορφώσουμε άποψη. Υπήρξε θαυμάσια συνεργασία και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτά τα δυόμιση χρόνια που είμαι επίτροπος για το πρίμα. Είναι το κυριότερο θέμα για το οποίο είμαι περήφανος κατά τα πρώτα δυόμιση αυτά χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθήσατε σε όλη την διάρκεια σε όλο το ταξίδι που κάναμε για να περάσει το πρίμα που ήταν ένα μακρύ ταξίδι αλλά τα καταφέραμε. Ευχαριστώ. Θέλω να σε ενημερώσω για τρία θέματα. Το πρώτο, που είναι νομίζω το κυριότερο, είναι η ενδιάμεση αξιολόγηση του Horizon 2020 και κατόπιν να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα εργασιών μας για το 18, 19 και 20 και το περαιτέρω πρόγραμμα για την καινοτομία που ο πρόεδρος ο πρόεδρός μας αποκάλεσε Horizon 2027 θα δούμε τι όνομα θα του δώσουμε και να μου κάνετε παρακαλώ και προτάσεις για το όνομά του. Και τα τρία αυτά θέματα, αξιολόγηση, πρόγραμμα εργασιών και το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, συνδέονται με την έκθεση Καμπεθών Ρουίθ για την αξιολόγηση του ορίζον 2020, που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά τη συζήτηση που κάναμε στην Ολομέλεια, μαζί σας. Καταλάβαμε ότι η έκθεση αυτή έχει παρόμοιες ιδέες με τις δικές μας για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, που είναι οι ευκαιρίες, που είναι οι δυσχέρειες. Άρα πολύ σημαντική συμβολή, κατά τη γνώμη μου, στην προετοιμασία του επομένου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας. Λοιπόν, τώρα, πώς πάει τώρα η ενδιάμεση αξιολόγηση. Είχαμε περίπου 3.500 απαντήσεις στη διαβούλευση που ξεκινήσαμε από 69 χώρες. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Και είχαμε και πάνω από 300 έγγραφα τοποθέτηση. Όταν είδα τα νούμερα για πρώτη φορά νόμιζα ότι είχε γίνει λάθος γιατί είναι τεράστια νούμερα. Και από παντού. Και εντός και εκτός Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ γνωστό παντού στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Τώρα, ορισμένα σημεία για το πώς ε, κατραίνω εγώ τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης και της αξιολόγησης. Πρώτον, Το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 θεωρείται ότι τα πάει καλά και είναι πολύ ενδιαφέρον για τους ενδιαφερόμενους και θα επιτύχει κατά πάσα πιθανότητα τους στόχους του. Άρα η αξιολόγηση των στόχων του 2020 εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να είναι πολύ επίκαιρη και στα πλαίσια των νέων παγκοσμίων προτεραιοτήτων ε, της Ένωσης, αλλά και για την επίτευξη των ε, βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Άρα τα πάμε καλά και συμβαδίζουμε με την πορεία εφαρμογής των ε, παγκοσμίων βιωσίμων στόχων. Και παράλληλα, αποδείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε και ευέλικτοι και με την κρίση του έμπολα, με την κρίση του ΖΙΚΑ και σε άλλες περιπτώσεις. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να δράσουμε με ευελιξία. Σήμερα Έχουμε λάβει για το Horizon 2020 πάνω από 145.000 προτάσεις. Καταλαβαίνετε πόση διοικητική στήριξη πρέπει να έχουμε για να τις αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Αν χρηματοδοτούσαμε όλες αυτές τις προτάσεις, θα χρειαζόμασταν 255 δις. Ακόμη και αν ήταν δηλαδή δυνατό, θα θέλαμε τόσα λεφτά. Αλλά δυστυχώ, η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμη και μερικές πολύ καλές προτάσεις. Χρηματοδοτούμε μία στις τέσσερι από τις ε, βέλτιστε Αυτό είναι κρίμα. Και αυτό πρέπει να είναι δίδαγμα και για το μέλλον. Τι θα γίνει, τι αποτέλεσμα έχει όταν έχεις τόσες καλές προτάσει και μπορεί να εφαρμόσεις μόνο τη μία στις τέσσερι. Το δεύτερο είναι συνεργασία. Και πολλά πρέπει να δούμε για το πώς ε, λειτουργεί η συνεργασία. Και ορισμένες επικρίσεις έχουν διατυπωθεί ότι δεν συνεργαζόμεθα όσο θα έπρεπε και όσο ήταν στο παρελθόν. Αλλά είναι παρόμοια η κατάσταση, όπως και στο 7ο πρόγραμμα. 75% της χρηματοδότησης πηγαίνει σε μέσα που ε, ευνοούν τη συνεργατική έρευνα. 75%. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στο ERC που είναι επιδοτήσεις ε, για μεμονωμένους ερευνητέ και επίσης το μέσο για τις μικρομεσαίες που είναι θαυμάσιο πιστεύω. Και θα σας πω, πάνω από μία στις πέντε δημοσιεύσεις βασίζονται σε συνεργασία του πανεπιστημιακού χώρου με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μία από τις σημαντικές αλλαγές που έχω διαπιστώσει στα πανεπιστήμια είναι ότι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο με την ε, οικονομία. Και εμείς παίξαμε γιατί ρόλο σε αυτό. Πολλές δημοσιεύσεις. Το είδα αυτό και όταν πήγα στην Ιρλανδία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η Ιρλανδία έχει ένα δίκτυ που δείχνει οι μελέτες και οι εργασίες που βασίζονται σε συνεργασία ε, αναφέρονται περισσότερο και από άλλους μετά. Πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν αυτή η συνεργασία. Και κάτι άλλο που είναι καταπληκτικό επίσης. Ότι συμμετέχουν οργανώσεις στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας από πάνω από 130 χώρες. Πολύ λίγα πιστεύω προγράμματα στον κόσμο έχουν τόσο ευρεία συμμετοχή. Μεγάλες χώρες επίσης. από όπου συμμετέχουν πολλοί. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί στον κόσμο. Τρίτον, το τρίτο μήνυμα από την αξιολόγηση μετά την ε, διαβούλευση είναι ότι το ορίζον 2020 θα επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων σε σχέση με το κόστος. Είναι πολύ βασικό να καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ απλό πρόγραμμα το 2020. Ελάχιστα γραφειοκρατικό. Από τα, λιγότερα, από τα λιγότερο γραφειοκρατικά προγράμματα στην Ευρώπη. Βεβαίω κάνουμε ένα δεύτερο ε, κύμα διαδικασιών απλούστευσης. Και όταν το ξεκινήσαμε, οι απαντήσεις που πήραμε είναι ότι το Horizon 2020 είναι πολύ απλούστερο από πολλά εθνικά προγράμματα. Νομίζω πως αυτό ήταν ε, επίτευγμα του Κοινοβουλίου. Εκεί αποφασίσατε ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, δύο ποσοστά χρηματοδότησης, ότι τα έμεσα έξοδα θα χρηματοδοτούνται κατά αποκοπή. Όλα αυτά συνέβαλαν σε αυτήν την ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων. Το τέταρτο μήνυμα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμη σταγόνα των ωκεανών. Εγώ το αποκαλώ ε, το πρόγραμμα του των 2-8%. Είμαστε το 8% των επενδύσεων στον τομέα στην Ευρώπη και 8% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Είναι ο ίδιος αριθμό, αλλά είναι δύο διαφορετικά, αναφέρονται σε δύο διαφορετικά μεγέθη. Και όταν ε, πρόσφατα συναντήθηκα με τον ε, πρόεδρο του NHS των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ρώτησα για τον ετήσιο προπολογισμό των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και μου είπε 30 δις το χρόνο. Εγώ νομίζω ότι έκανε λάθο. Δεν θεωρούσα ότι είναι, είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλο αυτό ο προπολογισμό. Μα τι καταδεικνύει αυτό. Χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν τόση ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο δικό μα ενωσιακό επίπεδο χρηματοδότηση. Είναι μόνο 8%. Σε χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάνω από 50%. Μικρό ποσοστό λοιπόν. και έχουμε και περιορισμένους πόρους σε σχέση με τον προπολογισμό της Ένωσης. Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει να το επανεξετάσουμε. Θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο για περισσότερες ε, πιστώσεις. Κάντε μου παρακαλώ ένα νόημα όταν θα πρέπει να τα τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ. Το πέμπτο που ήθελα να αναφέρω είναι επειδή εστιάζει στην ε, επιστημονική, οικονομική και κοινωνική επίπτωση, το ορίζον 2020 θα συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ολομέλεια, είχα την ευχαρίστηση για δεύτερη φορά την ίδια μέρα να είμαι στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε την έκθεση Λαμπατζόβα, Γιάλα Σέντερ για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και με χαρά διαπίστωσα ότι και η έκθεση αυτή αναγνωρίζει ότι χειριζόμεθα χρηστά τους πόρους μας. Άμα δείτε ότι για πρώτη φορά έχουμε τόσες εργασίες που παράγονται που μετά αναφέρονται τόσο πολύ σε άλλες εργασίες. Έχουμε ένα μητρό αυτών των αναφορών που δείχνει ότι είμαστε στο διπλάσιο του παγκοσμίου μέσου όρου. Αυτό αποδεικνύει όχι μόνο πως κάνουμε καλή χρήση των πόρων, αλλά είμαστε και αποτελεσματικοί σε αυτά που κάνουμε. Δεν είμαστε λοιπόν απλώς αποτελεσματικοί στη χρήση των πόρων. Και αν δείτε τι επίπτωση έχουν όλα αυτά στην οικονομία, και χθε είχα τη χαρά να είμαι στην Νορβηγία για ένα καταπληκτικό φεστιβάλ μουσικής και επιστήμης και ένας νομπελίστας μας είπε Κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη προέρχεται από την καινοτομία και την επιστήμη κατά πάνω από 60%. Για κάθε ευρώ διαπιστώσαμε που δίνουμε στα προγράμματά μας μπορείς να έχεις ε, αύξηση κατά 6 8% μέχρι το 2030. Βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη δουλειά μας και να σας πω τι πρέπει να βελτιώσουμε και να ακούσω και τη δική σας ε, αντίδραση. Πρέπει να βελτιώσουμε σε διάφορους τομείς. Ο πρώτος τομέας έχει να κάνει με το πόσο πολλοί υποβάλλουν προτάσεις. Θα θέλαμε άλλα 60 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουμε όλες τις προτάσεις που τώρα χρηματοδοτούνται μόνο κατά το 1 τέταρτο. Δηλαδή όλε τις πολύ καλές προτάσει ποιοτικέ. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε συμφωνώ με την πρότασή σας για τα 120 δις ευρώ. Σας συγχαίρω για το θάρρος σας. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε αυτή την υπερβολική υποβολή προτάσεων. Ίσως θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η υποβολή προτάσεων γίνεται, ε, συγγνώμη, οι υποβληθήσεις προτάσεις εξετάζονται σε δύο φάσεις για να μην συμμετέχουν πολύ στη δεύτερη φάση. Ο δεύτερος τομέας όπου εργαζόμεθα πάρα πολύ και μας έχετε βοηθήσει ιδιαίτερα και βλέπω πολλούς συναδέλφους που μας έχουν βοηθήσει εδώ παρόντες σήμερα για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των δυσχεριών που προκαλούν οι καινοτομίες Και ξέρω ότι είναι κάτι που το συζήτησε και το Συμβούλιο Καινοτομία και μας έχετε στηρίξει πολύ. Να δημιουργήσουμε τρόπους για να γίνονται, να προκύπτουν από τη βάση οι καινοτομίε. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Γιατί αλλιώ θα έχουμε πρόβλημα. Χθε μίλησα με μια εταιρεία που μας είπε ότι ήθελα να συμμετάσχουν στα προγράμματά μας και δεν μπορούσαν γιατί θεωρούν το υπερβολικά καινοτόμοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Το άτομο με τον οποίο συζήτησα είναι ένα άτομο που παράγει ηλεκτρισμό από τα φυτά. Από μια Ολλανδική εταιρεία που λέγεται Plant E. Αλλά επειδή εργαζόταν λοιπόν σε δύο τομείς, φυτολογία και ηλεκτρισμό, τους μπέρδεψε. Και το βασικό λοιπόν είναι να συμμετάσχει και η κοινωνία. Πρέπει η επιστήμη και η καινοτομία να είναι πιο στοχευμένες. Όταν ο Κέννεντι ανέφερε συγκεκριμένο στόχο, να βάλουμε, να πάει κάποιο στο φεγγάρι, να μπορέσει να πάει κάποιο στο φεγγάρι. Αυτό δεν ήταν απλώ ένα σύνθημα, βοήθησε να γίνει πιο στοχευμένη η έρευνα. Θυμάστε αυτόν τον επιστάτη που καθάριζε όταν πήγε στην NASA ο Κέννεντι και ο Κέννεντι τον ρώτησε, τι κάνει εδώ πέρα καθάρισε και είπε βοηθάω να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο εστιασμένη η προσέγγιση μας. Έτσι θα ευαισθητοποιούνται και θα συμμετέχουν περισσότερο οι επιστήμονες. Τώρα, συζητάμε το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2018-19-20. Συνεργαζόμεθα με όλες τις πλευρές και συνεργάζομαι και με τους συναδέλφους μου για να καθορίσουμε τις προτεραιότητες που τις ξέρετε, που τις αναφέρω πολύ συχνά αλλά η εργασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες και μάλιστα με καλό τρόπο. Και μετά νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τις χρηματοδοτήσεις των θεμάτων που θα επιλέξουμε. Και για το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο, το έχω πει επανειλημμένα, θέλουμε να υπάρχει αριστεία, ανοιχτό πνεύμα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτά θα πρέπει να είναι στο κέντρο των προγραμμάτων μας, είτε είναι το ένα το πρόγραμμα, είτε το ε, ορίζον 2027, να δούμε και ακούω και τις προτάσεις σας. Πρέπει να αιτιολογούμε πάντα την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων μας. Και γι' αυτό πρέπει να είναι ακριβώς. Άριστα τα προγράμματα πρέπει να είναι ανοιχτά και να έχουν επιπτώσεις παντού κοινωνικές για μια καλύτερη κοινωνία για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι το νέο αυτό πρόγραμμα, το ένατο, θα είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης και τεχνολογίας για μια καλύτερη επιστήμη, επιστήμης και καινοτομία για μια καλύτερη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είναι ιδιαίτερη αυτή η μέρα για σας, για μας. Μάλιστα υποδεχθήκαμε και έναν αρμόδιο από το γραφείο σας. Θα περάσουμε στη συζήτηση με πρώτους τους συντονιστές από, τους, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Έλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Εγώ θα έλεγα να πούμε να αναφερθούμε στο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα των 100 εκατομμυρίων. Γιατί δεν αναφερόμαστε στο μέλλον και ίσως 120 δισεκατομμύρια είναι ο καλός τίτλος για το νέο πρόγραμμα, αντί να αναφέρουμε μια ημερομηνία. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Τι γίνεται με την υπερβολική υποβολή ετήσεων. Μας εξηγήσετε τους λόγους. Τι θα γίνει όμως για το υπόλοιπο διάστημα. Θα αυξήσουμε το ποσοστό μήπως ή θα το κρατήσουμε μετάβλητο και θα παραπονιόμαστε ή θα χρειαστούν περισσότερα κονδύλια. Θα χρειαστούμε συγκεκριμένες απαντήσεις την επόμενη διετία. Δεύτερον, για το ευρύτερο πλαίσιο. Ε, Είπαμε ότι η σφραγίδα της αριστείας είναι ένα χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ε, τώρα ξεκινούμε συζητήσεις ε, για τα διαρθρωτική και άλλα ε, συναφή ταμεία και κάποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως της Δημιουργικής Ευρώπης. Ποιο είναι το ευρύτερο όμως πλαίσιο για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Επίσης, ε, συνοπτική διαδικασία για την καινοτομία. Ίσως ε, ε, θα μπορούσαμε να την θεωρήσουμε ως μία από τις τρεις βασικές προτεραιότητες και αυτή είναι η γνώμη και του κλάδου και ήταν πολύ θετική ανταπόκριση κυρίως από τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του προγράμματος. Θα διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός, θα είναι πλήρες πρόγραμμα ε, ή θα το αναλάβει η IC. Ποια, ποια είναι η προοπτική. Τέλος. Ποια είναι η αντίληψη του κοινού για το τι είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κβαντικό θα έλεγα σχέδιο ε, το πιο δημοφιλές που θα έχει απήχηση και στο κοινό και θα μπορέσουμε να το προβάλλουμε και από πολιτική άποψη και πραγματικά θα είναι ρηξιγέλευθο και ανατρεπτικό για τα μάτια του κοινού και θα μπορεί να το κατανοήσει ο απλός κόσμος και δεν θα είναι ένα περίπλοκο σχήμα διανοητικά, αλλά θα μπορέσει να φέρει τον κόσμο με ένα, μια, με ένα αντιληπτό όρο πιο κοντά στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη. Η κυρία Καμπεσόν Ρουή από του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για αυτά που είπε για το ένατο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Πολύ ενδιαφέρονται τα σχόλιά του και ευθυγραμμίζονται και με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω δύο γενικά σχόλια και δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις. Καταρχήν, ποια είναι η νέα πιθανή GTI για την υπερπροσφορά αυτή και θα έχουμε επιπλέον προϋπολογισμό από τα κράτη-μέλη. Και δεύτερη συγκεκριμένη ερώτηση δεν ξέρω αν ευσταθεί, ο Καναδάς όντως έδειξε ενδιαφέρον για να περιληφθεί στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Και ε, τι γνώμη έχετε για αυτό το άνοιγμα του προγράμματος προς τρίτες χώρες που ανάλογα με τη συμβολή του στο πρόγραμμα, με τη συνεισφορά του στο πρόγραμμα θα μπορούσαν να λάβουν και αυτές μέρος. Ε, ως προς τον προϋπολογισμό τώρα. Είπατε ότι ορίζοντας 2020 το, πρόγραμμα, το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που είναι πολύ άριθμες. Και το 80% είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα αύξηση του προπολογισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο το 1, το να φτάσουμε δηλαδή στα 120 δις. Και πέραν τη συνέργεια με τα διαρθρωτικά και άλλα ταμεία, η συμμετοχή των κρατών μελών έχει κέρια σημασία. Σκέφτεσαι κάποια μέτρα για να δώσετε ενάψματα στα κράτη-μέλη και να φτάσουν στο επιθυμητό 3% όλα όμως. Επίσης, μας είπατε ε, ποια ήταν τα πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης ε, για τον ορίζοντα 2020 και την ενδιάμεση αξιολόγηση. Και μας είπατε ότι ήταν πολλές οι συνεισφορές που λάβατε. Έχουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπονήσει μια έκθεση μετά από ακροάσεις, ε, ομάδες εργασίας, σεμινάρια. Μια έκθεση που συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία που χρειαζόμαστε και για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για να δώσουμε εμπιστοσύνη στο μέλλον. Αναφέρονται πολλά μέτρα στο, στην έκθεση αυτή. Ποια είναι η γνώμη σας. Πάντως είναι σημαντικό να σας στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το, 7 για το επόμενο, το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο, γιατί εμείς είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, οπότε πρέπει να, τύχετε και τις δικές μας υποστήριξης. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των φιλελευθέρων. Η κυρία Βίρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να πω τα εξή. Για το πρόγραμμα πλαίσιο, το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο, ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειε για να το κάνει πιο εύκολο και για να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Μιλάμε για 120 δισεκατομμύρια και δεν είναι μόνο θέμα επιθυμιών μας, αλλά είναι και θέμα αναγκών της Ευρώπης. Η αριστεία, το ανοιχτό πνεύμα και ο αντίκτυπος είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Και για τα διαθετικά ταμεία, όπως είπε η συνάδελφος ήδη, θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να συνδεθούν τα διαφορετικά ταμεία, η καινοτομία, η έρευνα και το Horizon 2020. Ε, να συνδεθούν με το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο. Προσβλέπουμε στην μελλοντική συνεργασία μαζί σας, όπως όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νταλούντε, εκ μέρους των Πρασίνων. Κύριε Νταλούντε, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την σημερινή σας επίσκεψη και για τη συζήτηση μαζί μας. Έχω ερωτήσεις για την κλιματική αλλαγή και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η αιτιολογική σκέψη 10 βάζει ένα στόχο 60% του προϋπολογισμού του 2020 που θα πρέπει να δίδεται στην ε, έρευνα για, την κλιματική αλλαγή και θα πρέπει ε, το 35% του υπολογισμού του Horizon να διατίθεται σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Αλλά στην αξιολόγηση την οποία έχει ενώπιον της η Επιτροπή φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις εναντί της επιτεύξης του στόχου. Βάσει τη συμφωνία του Παρισιού, μπορεί να δει κανείς ότι η τωρινή εξέλιξη δεν είναι αποδεκτή. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, τι θα κάνει η Επιτροπή για να διορθώσει την κατάσταση αυτή στα τελευταία χρόνια του τρέχοντος προγράμματος, ούτως ώστε να επιτύχουμε τελικά το στόχο. Και δεύτερον, είναι έτοιμη η Επιτροπή να προχωρήσει περισσότερο για το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο, ιδίω ε, εφόσον το Κοινοβούλιο στην τελευταία ολομέλεια ε, του ε, Στρασβούργου ε, ψήφισε υπέρ της χρηματοδότησης μέτρων για την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Άλλοι ομιλητές, η κυρία Κουντρίτσκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια ερώτηση προς τον Επίτροπο. Η συνάδελφος ε, μίλησε για, την, για το ψήφισμα που εγκρίναμε στις 13 Ιουνίου. Εδώ είμαι, κύριε Επίτροπε. Στο ψήφισμα, λοιπόν, της 13 ε, Ιουνίου... Εμ, εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από 520 ψήφους ε, συγκέντρωσε θετικές. Στο ψήφισμα μάλιστα αυτό επισημάναμε πολλά προβλήματα που διαπιστώσαμε στη λειτουργία του ορίζοντας 2020. Εσείς ε, τι προτείνετε για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα που επισημάναμε και εμείς στο ψηφισμά μας. Γιατί ε, μας προβληματίζει και περιμένουμε συγκεκριμένες ε, και αυτές απαντήσεις. γιατί μας μιλήσατε για την ανταγωνιστικότητα και τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά σήμερα ε, δημοσιεύθηκε το European Innovation Scoreboard, όπου αναφέρεται ότι η Ευρώπη είναι λιγότερα καινοτόμα από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την ε, Νότια Κορέα και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό δείχνει ε, ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αξιολόγησης για την Καινοτομία. Ε, κάτι που δείχνει ότι μπορεί να έχουμε πολλές δημοσιεύσεις ε, και συζητήσεις για την καινοτομία, αλλά στην πράξη τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης καινοτομίας και της υστέρησης. Γιατί θέλουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουμε ε, δύναμη παγκόσμια στην καινοτομία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Και θα πρέπει να μεριμνήσουμε σε τα πιο δύσκολα προγράμματα και σχέδια να χρηματοδοτηθούν. Συνεχώς λοιπόν προβληματίζομαι για αυτό το θέμα. Πώς θα διαμορφωθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία, ποιο θα είναι το χαρτοφυλάκι αυτού του Συμβουλίου, τι προϋπολογισμό θα διαθέτει, πότε επιτέλους θα θεσπιστεί και θα αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι ένας τέτοιος νέος θεσμικός φορέας θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δραστηριότητές της ως προς την καινοτομία. Ελπίζω να μας ενημερώσετε όσον πω για τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Κουντρίτσκα. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Πολ Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι μέλος Επιτροπής Προϋπολογισμών και πάντα τίθεται το θέμα, όταν συζητάμε το πολιετές πρόγραμμα πλαίσιο, πώς θα επιλέξουμε τους σωστούς τρόπους, ε, γιατί θα παίξει ρόλο και το Brexit. Πώς θα εξέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τι τρόπο θα συμμετάσχει ενδεχομένως στο μέλλον. Και σε τι βαθμό θα χρειαστούν ε, αυξήσει στον προπολογισμό μας. Νομίζω ότι κάθε περίοδο θα έπρεπε να απαιτούμε το διπλασιασμό του προπολογισμού μας. Γιατί μετά βέβαια οι υπουργοί θέλουν να κάνουν ε, περικοπές. Αυτή είναι η διαδικασία. Εμείς ζητάμε περισσότερα και αυτοί αποφασίζουν περικοπές. Επί της ουσίας θα ήθελα να μάθω τι θα γίνει με την ε, γλωσσική τεχνολογία. Τις τελευταίες, τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει ραγδαίες εξελίξεις. Και κάτι άλλο που το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί για τα κούκι, τα ηλεκτρονικά μπισκοτάκια και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται τώρα στα δίκτυα. Την ε, την τεχνητή νοημοσύνη και ποια προγράμματα θα τα βοηθήσουν όλα αυτά ούτως ώστε να εστιάσουμε κυρίως σε αυτόν τον ε, ψηφιακό κόσμο και το τρίτο οι μπαταρίες παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο οι μπαταρίες οι ιόντων λιθίου ξαφνικά παίρνουν φωτιά τι θα γίνει εάν ένα αυτοκίνητο, για παράδειγμα, παρκάρει σε ένα υπόγειο γκαράζ με 400 κιλά τέτοιας μπαταρίας και πάρει φωτιά και δεν μπορούμε να τη σβήσουμε. Τι θα γίνει αν, αν καεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, να θέσουμε θέματα, να δούμε δηλαδή για παράδειγμα ποια είναι η ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας, ε, προς τα που πρέπει να προσανατολίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ. Κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, εν μέσω κρίσης, όπως ο πολιτισμός, η καινοτομία είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που περικόπτεται. Γιατί δεν έχει άμεση απόδοση, άμεση επιστροφή και στην οικονομία δυστυχώς θέλουμε αμέσως αποτελέσματα ε, και γι' αυτό ο πολιτισμός και η καινοτομία βγαίνουν χαμένοι. Αλλά αυτό που μας λείπει δεν είναι οι ιδέες, τα μέσα είναι που μας λείπουν. Γιατί όταν αναφερθήκατε στην κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν ε, ε Δείτε τι γίνεται στη Silicon Valley και βλέπετε ότι πολλά εργαστήρια ευρωπαϊκά βρίσκονται εκεί στην Silicon Valley γιατί εκεί έχουν ελευκό επιταγή ε, και έχουν όλα τα μέσα για να φέρουν σε πέρα στις έρευνές τους. Ναι λοιπόν λέμε στην έρευνα, αλλά για ποιο λόγο και για ποιον. Είναι σημαντικό να απαντήσουμε και σε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί και για ποιον. Μιλήσαμε για την ενεργειακή πολιτική, την αηφόρο ανάπτυξη, τις νέες ενέργειες και αυτή αυτό είναι προτεραιότητα, ο άξονας προτεραιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξυπηρετεί του πολίτε και τον πλανήτη. Εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει πολυάριθμες έρευνε για τι ΑΠΕ, για, τις, ε, ε, ε, για την αιωλική ενέργεια, για κάποιες τεχνικέ που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια που, ανα, που προορίζονται για τις περιφερειακές ζώνες ε, χρησιμοποιώντας ε, τη, την δύναμη της θάλασσας και των κυμάτων και τη διαφορά θερμοκρασίας ανάλογα στα ανώτερα και στα βαθύτερα επίπεδα της ε, ε θάλασσας. Υπάρχουν πρωτότυπα, αλλά δυστυχώς σκουριάζουν, βρίσκονται σε κάποια συρτάρια, γιατί δεν έχουμε κονδύλια να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Και για την COP21 θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη φιλοδοξία για να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς αύξηση θερμοκρασίας. Αλλά ε, οι περιφερειακές ζώνες είναι διπλά καταδικασμένες γιατί είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν μαζούτ ε, άνθρακα για την ενέργειά τους, τις πιο ρυπογόνες, δηλαδή πρώτες σύλλες, και επίσης ε, είναι υποχρεωμένες να εισάγουν μηχανήματα που είναι πολύ ακριβά. Οπότε είναι διπλά θύματα οι πιο απόμακρες περιοχές και οι περιφερειακές ζώνες. Πώς λοιπόν ε, θα απελευθερώσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Μπορεί να έχουμε έναν επίτροπο που δίνει μάχη και λέει είναι σημαντική καινοτομία, θα πρέπει να τη στηρίξουμε και από την άλλη να έχουμε άλλο επίτροπο που λέει Α, το Ταμείο είναι μείον, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την καινοτομία και την έρευνα. Θα πρέπει να είμαστε συνεπεί. Μπορείτε λοιπόν να τα αποδεσμεύσετε αυτά ώστε όταν χρηματοδοτούμε την καινοτομία, ε, όταν προωθούμε την καινοτομία να την συνοδεύουμε και με απαραίτητα κονδύλια για την απαραίτητη βιομηχάνηση και με αρκετά προσιτές τιμές ώστε να υποφεληθούν όλοι. Ευχαριστώ. Um, thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Νίβλα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρία πολύ σύντομα ερωτήματα. Καταρχήν, όσον αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση. Ε, το μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις νομίζω ότι έγινε πολύ καλά αποδεκτό και θα μπορούσατε να πείτε κάτι παραπάνω. Μια δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό βασική έρευνα. Γνωρίζετε σε τι βαθμό προκύπτουν καινοτομίες από τη βασική έρευνα. Και μια τρίτη και πιο σημαντική ερώτηση αφορά την εποχή μετά το Horizon 2020, ε, το νέο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα έχει το τίτλο, «Καινοτομία για καλύτερη κοινωνία». Έχετε κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί της Επιτροπής για την προετοιμασία του ενάτου προγράμματος πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ντανίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας για το διάλογο αυτό, όπως πάντοτε μας επισκέπτεστε. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Ήταν ιδιαίτερα ενημερωτική. Δυστυχώς, όσοι γνωρίζουν πραγματικά το δυναμικό των κονδυλίων και της χρηματοδότησης για το Horizon 2020 είναι πολύ λίγη και αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση θα είναι πολύ χρήσιμη για μας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποια ερωτήματα τα οποία μας ανησυχούν για τα θέματα αυτά. Ανησυχούμε διότι παρά τις ε, προσπάθειές μας να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στον τομέα των μεταφορών και επομένως υπονομεύονται αυτές οι προσπάθειες. Από όσο γνωρίζω, ο κύριος λόγος είναι ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν έχει πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνολογία για ηλεκτρικούς κινητήρες οχημάτων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για απόσταση πάνω από 300 μίλια. Ε, προβλέπει η Επιτροπή κάποια έρευνα στον τομέα αυτό που θα δημιουργήσει ε, μια νέα εποχή γιατί όσο δεν δίνουμε κίνητρα δεν θα υπάρχει και αποτέλεσμα. Εάν δεν βιαστούμε βλέπουμε ότι η Κίνα κάνει τεράστιες πρόοδους και παράγει ηλεκτρικά οχήματα και ηλεκτρικά λεωφορεία. Στην Ευρώπη είναι πολύ αργή η πρόοδος στον τομέα αυτό. Αυτό το προκαλούν και οι κατασκευαστές στον τομέα αυτό που δεν δίδουν τα απαραίτητα μέσα στους χρήστες που θέλουν μεν ηλεκτρικά οχήματα αλλά δεν έχουν τρόπο να τα φορτίσουν. Ε, ένα άλλο θέμα τώρα, η ιατρική έρευνα. Εδώ έχουμε ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ. Πολιτείες. θα πρέπει να επιτρέπουμε σε όσο δυνατόν λιγότερους ε, πολίτες να θέλουν να πάνε ε, στις ΗΠΑ για ε, θεραπεία. Βλέπουμε ότι οι ασθενείς θέλουν να πάνε στις ΗΠΑ γιατί είναι πολύ προηγμένες οι τεχνικές και η θεραπεία και στην Ευρώπη δεν έχουμε πρόσβαση σε τόσο προηγμένη θεραπεία όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα συναντήθηκα με μία ένωση ασθενών που ε, πάσχουν από καρκίνο του στομάχου και μου είπαν ότι δίνονται τόσο λίγα κονδύλια για έρευνα που ακόμη και οι εξειδικευμένες κλινικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη και τα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα δεν καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και βάσει των στατιστικών στοιχείων δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Ξέρω ότι δεν είναι απόλυτα δική σας αρμοδιότητα αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα κάποια σχόλια και για την ιατρική έρευνα. Για πολλούς από εμάς είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Επιτροπέ πολύ σωστά λέτε ότι θα πρέπει να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στην έρευνα και στην ε, καινοτομία. Ο κύριος Σέλλερ θέλει ένα σύνθημα και ίσως αυτό που ακούσαμε σε μία διάσκεψη, το να φτάσουμε σε ποσοστά 0 το 2050, ε, είναι ένα σύνθημα που μπορεί να μας οδηγήσει σε πρόοδο σε πολλούς τομείς. Αυτό αφορά και την τεχνολογία, αλλά υπό κάποια έννοια αφορά και τα δίκτυα και την κοινωνιολογική προσέγγιση, τη ζωή των πόλεων κλπ. Υπάρχει το πρόγραμμα για την ενεργειακή εξυπνάδα στην Ευρώπη και νομίζω ότι δεν έχει την επαρκή ορατότητα αυτό το πρόγραμμα. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορείτε το, στην επόμενη περίοδο να έχετε περισσότερο ήπιες πολιτικές που θα αφορούν τις μεταφορές, την αλλαγή του κλίματος, αλλά να έχουν ορατότητα όλα αυτά. στην αρχή ήταν πολύ ε, έντονα όλα αυτά τα θέματα, αλλά χάσαμε σιγά σιγά ε, όλα αυτά τα θέματα από ε, τα μάτια μας και πρέπει να τα επαναφέρουμε. Το επόμενο θέμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα. Έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Από παγκόσμιος ηγέτης κινδυνεύουμε να χάσουμε τη θέση μας. Και αυτό αναδεικνύεται ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη, θα χάσουμε μεγάλο βαθμό της παραγωγής, 45% της παραγωγής ε, ηλεκτρικών οχημάτων. Χρειαζόμαστε ε, υποστήριξη όσον αφορά τις εταιρείες ενέργειας χρειαζόμαστε υποστήριξη και στον τομέα των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αν εμείς κάνουμε ε, επένδυση 5 δισεκατομμυρίων, βλέπουμε ότι οι Κινέζοι κάνουν πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις. Ποια είναι η κρίσιμη μάζα που θα μπορούσε να μας δώσει το προβάδισμα των ανταγωνιστών μας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σε σχέση με τα όσα γίνονται στην Κίνα τι μπορούμε να διδαχθούμε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι η κυρία Μόλντε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλά υπόθηκαν. Να αναφερθώ σε κάποια άλλα. συζητούσαμε μία οργάνωση έρευνας ε, κατά του καρκίνου. Και ορισμένοι μου είπαν ότι υπάρχει έρευνα, αλλά ο καθένας ε, στη γωνιά του δεν υπάρχει αρκετή σύνδεση και συνεργασία. Αν υπήρχε συντονισμός, θα μπορούσαν να έχουν πολύ περισσότερα αποτελέσματα από αυτές τις μεμονωμένες προσπάθειες. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία. Και αυτό με φέρνει και σε κάτι άλλο. Πώς θα ενημερώνουμε καλύτερα και τους πολίτε για αυτά που κάνουμε. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο και πιο αποτελεσματικά για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όχι για τα προγράμματα έρευνας, αλλά για το τι επιτυγχάνουν. Να, αυτή η θεραπεία αναπτύχθηκε, αυτή η θεραπεία άρχισε να εφαρμόζεται, αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είχε η έρευνα. Τα επιτεύγματα. Είπατε ότι χρηματοδοτείται μόνο 25% από τα πολύ καλά προγράμματα που προτείνονται. Τι είστε το θέμα, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε απογοήτευση. Δεν θα ε, υποβάλουν πια προγράμματα οι άνθρωποι. Ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να να χρηματοδοτούμε προγράμματα από όλες τις χώρες της Ένωσης, όχι μόνο από λίγες. Εδώ και η επιστήμη των πολιτών. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και κάτι άλλο που ήταν στη θαυμάσια έκθεση της Σολεδάδ που ψήφισαμε την επόμενη εβδομάδα. Να συμμετάσχει όσο περισσότερο και για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται η Βρετανία στα προγράμματα αυτά. Ξέρετε και έχω πει επανειλημμένα πόσο διαφωνώ με τον Brexit. Ό,τι Brexit και αν προκύψει, νομίζω ότι θα ήταν ε, αμοιβαία αποφελές να συμμετέχει όσο γίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει και να συμμετέχει και στη χρηματοδότηση, στον προπολογισμό. Να συμμετέχει λοιπόν και από τις δύο απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ρόλ. Κύριε Επίτροπο Ρόιλ, θα σας εκπλήξει. Δεν θα αναφερθώ σε ένα δικό μου θέμα, γιατί ο καθένας έχει αυτό που τον ε, ενδιαφέρει περισσότερο. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπατε ότι είπατε ότι μέχρι στιγμής ήταν ε, πολύ θετική η εφαρμογή του προγράμματος 2020. Οπότε τίθεται το ερώτημα τι θα πρέπει να αλλάξει. Όταν αποφασίζουμε για νέα πλαίσια θα πρέπει να έχουμε νέα ονόματα και νέες ιδέες. Το βασικό δεν είναι ότι αυτό που πάει καλά να το συνεχίσουμε απλώς να το χρηματοδοτήσουμε περισσότερο. Για μένα αυτό είναι το βασικό περισσότεροι πόροι, περισσότερες πιστώσεις. Εντάξει, αν κάποιος θέλει κάτι να αλλάξει, να μας πει. Ευχαριστώ να το ακούσω, αλλά το βασικό μας καθήκον είναι το άλλον. Δεν χρειαζόμαστε κάθε φορά νέες ιδέες και νέα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρία Grazie, Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Λυπάμαι, δεν πρόλαβα να ακούσω την παρουσίασή σας γιατί είχα μια πολύ σημαντική αντιπροσωπεία και μια συνάντηση εργασίας με συναδέλφους, με κάποιους ε, συμπατριώτες μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε οι προσπάθειές μας ε, να μην μείνουν ε, στη μέση και να καταλήξουν σε κάποια αποτελέσματα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Καταρχήν έχουμε θετήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση Καμπεσόν. Οι συστάσεις της έκθεσης Καμπεσόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνείτε ή όχι, θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στις προσπάθειες επιλογής των προτεραιοτήτων, ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Όταν αναλαμβάνουμε νέα προγράμματα, ποιος θα αποφασίσει για τους εμπειρογνώμονες και ούτω καθεξής. Θα ακούσετε τα, τις αιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλήσαμε για την εναλλακτική ενέργεια, την υγεία. Δεν θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάποιο λόγο στην επιλογή των προγραμμάτων για να αποφευθεί η υπερβολική διάχυση. Επίσης, αναφέρθηκε το Συμβούλιο Καινοτομίας. Ε, πώς ε, ξεκίνησε Ε, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι και το δικό μας έργο λαμβάνεται υπόψη και τροφοδοτεί τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχουμε υποβάλει πολλοί άριθμες προτάσεις. Θα πρέπει να τις δούμε να εφαρμόζονται κιόλα. γιατί έχουμε πολύ συχνά ενδιαφέρουσε και καρποφόρες συζητήσεις, αλλά δεν θα ήθελα να μένουμε στις συζητήσεις. Θα, ε, θέλω να έχουμε και λόγο στην επιλογή των προτεραιοτήτων. Είμαστε όντως ε, ενεργοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ήρθε η ώρα για βελτίωση της αλληλεπίδρασής μας και της επαφής μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Ματίας εκ μέρους της ΓΚΟΕ, τελευταία ομιλήτρια, με σχόλια και ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες ανησυχίες που έχω για κάποια σημεία του ορίζοντας 2020, ε, κυρίως ε, της χρηματοδότησης. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τις θεματικές ενότητες. Εγώ δεν προβληματίζομαι τόσο για τις θεματικές ενότητες, όσο για τους τομείς ε, γνώσης που θα χρηματοδοτηθούν από τον ορίζοντα 2020. Αυξήθηκαν οι δημοσιονομικές ικανότητες και τα κονδύλια για την καινοτομία, πολύ θετικό αυτό, αλλά όπως ξέρετε και το έχω πει επανειλημμένως, δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία αν αφήσουμε κατά μέρους ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αν δεν τροφοδοτήσουμε την βασική έρευνα, γιατί έτσι θα χαθεί η βάση και το υλικό για την καινοτομία. Και υπάρχουν σε ε, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του, πληθυσμού, του προϋπολογισμού να αναφέρεται στην καινοτομία. Αλλά τι γίνεται με την βασική έρευνα. Το ε, Ευρωπαϊκό Κέντρο καινοτομία ε, δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. γιατί και για τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες θα πρέπει να ξέρουμε τι χαρακτηριστικά έχουν οι κοινωνίες μας για να υιοθετήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές. Και γνωρίζουμε και όσοι ήμασταν ήδη ευρωβουλευτές ότι δυστυχώς ε, ε, ελάχιστα ελήφθηκαν υπόψη τον ορίζοντα 2020 παρά λίγο να μείνουν και εκτός ε, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Για τα ερευνητικά κονδύλια, τι γίνεται με άλλους τομείς, πώς χρηματοδοτούν την αμυντική πολιτική τα ερευνητικά κονδύλια, γιατί όλοι θέλουμε να αυξηθεί ο προπολογισμό, αλλά να μην αφιερωθούν ε, κονδύλια της έρευνας για άλλους σκοπούς. Για την άμυνα, για παράδειγμα. Δεν θα ήταν σωστό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο κανένα συνάδελφο να ζητά το λόγο. Μια σύντομη παρατήρηση ρώτησα για τον προγραμματισμό και τα λοιπά προγράμματα. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών, όπως είπε ο κύριος Τούρμες, θα εφοδιαστεί με ένα νέο όργανο για τις νέες τεχνολογίες. Αλλά και αυτό το εργαλείο είναι ξέχωρο, απομονωμένο. Τώρα ελήφθη η απόφαση ε, να έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για χαλιβουργίες ε, χωρίς ε, εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα. Και μάλιστα προβλέφθηκαν 500 εκατομμύρια. Τα 300 αφορούν το τεχνικό τμήμα και ακούσαμε ότι θα, αναφερ... θα χρηματοδοτήσουν άλλα θέματα, όχι την τεχνολογία. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε ένα πρόγραμμα για τον άνθρακα και το χάλιβα και άλλα 5-6 προγράμματα. Έχουμε το Ταμείο για την Εμπορία Εκπομπών. Θέλουμε να επιτύχουμε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, όπως είναι μια χαλιβουργία χωρίς, χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και πάλι διαπιστώνουμε ότι είναι κατακαιρματισμένη η χρηματοδότηση. Κύριε Κόχλησεκ, δεν θέλετε να λάβετε το λόγο πριν την κυρία Μα... Ματίας. Δεν θέλετε να κάθετε μπροστά της. Α, e, ε, Πραγματικά δεν θέλω να φύγω. Έχω τέσσερις ε, ε, σύντομες παρατηρήσεις. Ποια είναι τα μελλοντικά μας προβλήματα. Τι πορεία θα πάρει τεχνολογία. Το πρωί μιλήσαμε για πολλά και διάφορα θέματα και κατά τη γνώμη μου ε, μερικοί συνάδελφοι δεν κατάλαβαν ε, ότι η ολική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά, μερικές φορές ε, αποσταθεροποιούν το δίκτυο. Και είναι σημαντικό να έχουμε σταθερότητα του δικτύου για την ε, εύρυθμη λειτουργία ε, της, του δικτύου. Και είπα και το πρωί ότι οι Γερμανοί βρήκαν τη λύση αλλά και θα πρέπει να τους μιμηθούμε γιατί δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη να βρούμε ισορροπία μεταξύ όλων των τμήματων του δικτύου ιδιαίτερα για τι ΑΠΕ. Επίση, το θέμα των κλιματικών αλλαγών και του περιβάλλοντος είναι επίσημα σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Ε, θυμάστε πριν από τρία χρόνια δεν είχατε την ακρόαση, είχαμε το, δεν είχαμε τόσο εκτενή συζήτηση όσο σήμερα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πάντοτε χαίρομαι να έχω τόσες πολλές ερωτήσεις. Ε, ξεκινώ με τον κύριο Κρίσιαν Έλε. Νομίζω ότι ε, έχει δίκιο και συμφωνώ με τον αριθμό που προτείνεται τα 120 δισεκατομμύρια. Είναι όντως μεγάλο το ποσό, ιδίως ε, στις δύσκολες εποχές που έρχονται. Με ρώτησε ο κύριος Έλα και για το θέμα των του υπερβολικά μεγάλου αριθμού υποβολής αιτήσεων. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό όταν έχουμε περιορισμένο προϋπολογισμό, γιατί αν δεν έχουμε περισσότερα χρήματα, δεν έχουμε τη βάση για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο στη διαδικασία, να μην έχουμε απώλεια χρόνου σε δύο στάδια της διαδικασίας. Αν κάποιος περνάει από το πρώτο στάδιο και αποτυγχάνει στο δεύτερο στάδιο, να δούμε πώς θα μπορούσαμε ε, να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχία στο δεύτερο στάδιο, να είναι σαφέστερη η διαδικασία, να είναι η προκήρυξη σαφέστερη, να εξηγήσουμε καλύτερα τι ακριβώς θέλουμε, ώστε να μην χάνουν το χρόνο τους, εάν δεν είναι για αυτούς ε, η συγκεκριμένη προκήρυξη. Δεν μπορούμε να λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα του προπολογισμού. δεν έχουμε τα χρήματα για να το καλύψουμε όλο, αλλά μπορούμε στη διαδικασία των δύο σταδίων να προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε τη διαδικασία. Άλλη μια σημαντική ερώτηση του κυρίου Έλλερ αφορούσε την ταχεία διαδικασία για την καινοτομία. Και από άλλους συναδέλφους προέκυψε αντίστοιχο ερώτημα υπό διαφορετική μορφή υπάρχει μεγάλη κατάτμηση και προγραμμάτων και ονομάτων. Μερικά είναι πολύ επιτυχημένο, όπως αυτό το πρόγραμμα της ε, ταχείας ε, πορείας προς την καινοτομία. Και όπως είπα υπάρχει και το θέμα της καινοτομίας και της καινοτομίας που δημιουργεί διασπάσεις και τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε αυτή την γενική ιδέα που θα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ε, συνολικά. Και το βλέπω όταν έχουμε επαφή με το κοινό και το έλεγα και στους συναδέλφους στην Επιτροπή σήμερα ότι με όλα τα ονόματα που έχουμε για τα διάφορα προγράμματα ο κόσμος ε, χάνεται. Και ίσως το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των ονομάτων για να έχουμε ένα σήμα κατά να έχουμε ένα όνομα που θα είναι το όνομα που θα αναγνωρίζουν οι πολίτες ως πολιτική καινοτομία για την Ευρώπη. Και το πρόγραμμα που αναφέρατε τη ταχεία οδού προς την καινοτομία είναι το Fast Track, είναι ένα από τα αναγνωρίσιμα προγράμματα η αντίληψη που έχει λοιπόν ο πολίτης είναι σημαντική. Μερικές φορές δεν ξέρουν τι θα έπρεπε να κάνουν, που θα έπρεπε να απευθυνθούν και εδώ θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και γι' αυτό η ε, δέσμη μέτρων κάτω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία νομίζω θα βοηθήσει. Επίσης η σφραγίδα αριστείας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και στο ένα το πρόγραμμα πλαίσιο ε, θα δουλέψουμε με διαφορετικό τρόπο με τα διαρθωτικά ταμεία και ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητές μας και αν με ρωτήσετε ποιε είναι οι προτεραιότητές μα για τον ορίζοντα 2020, θα σα πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ευθυγραμμιστούμε με τι προτεραιότητε των Διευθυντικών ταμείων ε, για τι επιστήμε και την καινοτομία. Θα δούμε τι κονδύλια έχουμε και πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τις δράσεις μας, τουλάχιστον για θέματα προτεραιοτήτων. Αυτή είναι η γενικότερη ιδέα νομίζω. Και θα μιλήσω ισπανικά στη συνέχεια. Η κυρία Καβεθόν Ρουίθ με ρώτησε για το Καναδά. Εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση. για συζητήσεις με τον Καναδά για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Horizon 2020. Είναι σημαντικός σύμμαχος ο Καναδάς αλλά από όσο ξέρω δεν είμαστε σε συζητήσεις με τον Καναδά. Αλλά είναι σημαντικό σύμμαχος ε, του προγράμματος. Όπως και άλλοι που δεν συμμετέχουν αλλά με τους οποίους συνεργαζόμεθα. Για τους ε, υπερυπολογιστές GPI GTI Δεν έχω απαντήσει να σας δώσω. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον ε, κάποιες προτάσεις για το θέμα αυτό. Αν υπάρξουν ε, προγράμματα για τους ε, υπολογιστές σε πολύ μεγάλο δυνατοτήτων, στο ένα το πρόγραμμα πλαίσιο θα το δούμε. Για τον προϋπολογισμό. Αν θέλει η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρα στην τεχνολογία και την επιστήμη και να δημιουργήσουμε και θέσει απασχόληση, τότε πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί ο προπολογισμό μα. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται ούτε από εσά ούτε από μένα. Δυστυχώ. Και εμεί και εσεί το θέλουμε, αλλά το βασικό είναι και τα κράτη-μέλη να το θέλουν. Άρα θα είναι δύσκολο να τους πείσουμε ότι χωρίς επιστήμη, χωρίς τεχνολογία δεν έχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ανάπτυξη και χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει απασχόληση. Τώρα έχουμε την ερώτηση της κυρίας Βρίνκα. Αναφερθήκατε στο ένα το πρόγραμμα πλαίσιο. και τι αλλαγές θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Και αναφερθήκατε και στο θέμα της συνεργασίας με τα διατροτικά ταμεία. Ναι, είναι ουσιώδες. Βεβαίως, αυτή η σφραγίδα, το πιστοποιητικό αριστείας, ε, ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να εργαστούμε μαζί με τα, με τα διατροτικά ταμεία, γιατί έχουμε παρόμοιες προτεραιότητες. Επίσης ε, ε, μιλήσατε για τις διαφορές μεταξύ καινοτομίας και έρευνας. Αλλά δεν υπάρχει πάντα αυτή η διαφορά ανάμεσα στη βασική έρευνα και την τεχνολογία. Εγώ έχω δει πολλά θετικά αποτελέσματα από τη βασική έρευνα που καταλήγουν μετά σε καινοτομίες. Και έχω δει και πολλούς επιστήμονες που έχουν εργαστεί στον τομέα της καινοτομία και που μετά περνάνε στη βασική έρευνα. Ευχαριστώ πάντως για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Νταλούντε έχει δίκιο. Είμαστε στο 27% είπατε και ο στόχος μας είναι το 35% για την κλιματική δράση. και τα άλλα νούμερα που αναφέρατε. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, στο πρόγραμμα εργασιών για το 18-19-20, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να τα ιεραρχήσω, αλλά θα επιχειρήσω να τους πείσω ότι πρέπει να τα λύσουμε όλα αυτά. Και έχουμε τρία χρόνια. Αλλά το γεγονός ότι δεν επιτυχάνουμε τους στόχους ε, δεν είναι θετικό. για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ε, έχουμε μία προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν συνεισφέρει τα θέματα βιωσιμότητα και κλιματική δράση, αλλά δεν συνυπολογίζονται γιατί προέρχονται από το ERC. Δεν είχαν ονομαστεί προγράμματα για την κλιματική αλλαγή, αλλά ήταν στην ουσία, άρα πρέπει να δούμε πώς αξιολογούμε ορισμένα από τα έργα και πρέπει να τα παρουσιάσουμε με πλέον ορατό τρόπο. Προς την κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα. Θέλω καταρχήν να πω ότι ευχαριστούμε που αναφέρατε το θέμα της ε, βαθμολογίας της ε, καινοτομίας. Το scoreboard δείχνει ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουμε ακόμη μεγάλη πορεία μπροστά μας και οι διαφορές που βλέπουμε μεταξύ αυτών που κάνουμε εδώ και αυτών που γίνονται σε άλλες περιοχές του κόσμου οφείλονται στο ότι επενδύουμε λιγότερο εδώ από ότι επενδύουν σε άλλες χώρες. Και βλέπετε ότι στην Κίνα επενδύουν κάθε χρόνο και περισσότερο. Το βλέπετε και στην Νότια Κορέα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μία από τις μεγάλες διαφορές είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας στις χώρες αυτές επενδύει περισσότερο από ό,τι εδώ στην Ευρώπη. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε αυτό το Ταμείο των Ταμείων για την Ευρώπη, αυτό το Fund of Funds, για να προσελκύσουμε περισσότερα κονδύλια από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις. Εάν δεν προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Άλλες ερωτήσεις από άλλους βουλευτές αφορούσαν ένα άλλο θέμα για τους νέους επιχειρηματίες και προσπάθησα σε κάποιες συζητήσεις με νέους επιχειρηματίες ε, να τους πω τι θα μπορούσε να ε, ορίσει το EIC. Τους είπα ότι πρέπει να έχουμε ε, κάτι το οποίο θα είναι ορατό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας πρέπει να είναι ορατό. Και θα πρέπει, επειδή ε, εμφανιζόμαστε μέσω αυτού του μέσου, να θέλουν να επενδύσουν σε εμά ε, τα επενδυτικά κεφάλαια. Και θέλουμε κάτι το οποίο θα είναι σταθερό και θα έχει μια ε, συνολική εικόνα ισχυρή. Προσπαθούμε λοιπόν να αλλάξουμε και στο μέσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τις προκηρύξεις μας. Θα γίνονται, προκηρύ... γίνονται προκηρύξεις χωρίς ε, να λέμε αν θα είναι για τη βιολογία ή για άλλο τομέα ε, και βλέπουμε πώς θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και θα κρίνουμε αντιστοίχω. Επίσης, μέσω συνεντεύξεων μπορούμε να εντοπίσουμε ενδιαφέρουσε ιδέε. Αυτό λένε ε, όσοι επενδύουν σε καινοτόμε ιδέε. Λένε ότι ε, κάποιος ε, που είναι επικεντρωμένος ε, σε μία ιδέα, ακόμη και αν υπάρχουν αδυναμίες, ε, μπορεί να κάνει την ιδέα του να δουλέψει. Ακόμη και με μια λιγότερη καλή, λιγότερα καλή ιδέα, κάποιος που έχει τον ενθουσιασμό και τα κίνητρα μπορεί να οδηγήσει την ιδέα ψηλά, γιατί θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να καινοτομήσουν με ό,τι υλικό έχουν στη διάθεσή τους. Και γι' αυτό η καινοτομία θα συμπεριλάβει και μια διαδικασία συνεντεύξεων. Και προς την κυρία Τόγια, θέλω να πω ότι αυτή η ιδέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και μπορώ να το πω γιατί έχω κάνει αρκετές συναντήσεις και με ευρωβουλευτές και οι περισσότεροι ευρωβουλευτές ε, έχουν ιδέες και θέλουν να συμμετάσχουν περισσότερο. Και όταν συμμετέχετε σε σχετικές συναντήσεις πάντοτε έχετε πολύ σημαντική συνεισφορά. Θα φροντίσω λοιπόν, κυρία Τόγια, να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα φροντίσω να είναι γνωστό ότι κάνουμε τέτοιες συναντήσεις. Και προς τον κύριο Ρούμπι θέλω να πω όσον αφορά τις επιπτώσεις του Brexit και το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω προς το παρόν. Λυπούμε για αυτό που συμβαίνει, έχω εκφράσει τη γνώμη μου, αλλά τώρα από την έκφραση της γνώμης μου πρέπει να περάσουμε σε συγκεκριμένε πράξει. Μιλήσατε και για το θέμα των γλωσσικών τεχνολογιών και των αλγορίθμων ε, και ε, του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ έχουμε μια πολιτική επιλογή. Εάν θέλουμε να μας αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη ή αν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να επαυξήσει τη δική μας νοημοσύνη. Αυτή είναι η επιλογή μας. Εάν σωστά επιλέξουμε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Τώρα βλέπουμε αυτό το νέφος ε, της επιστήμης και πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτό το νέφος. Δηλαδή μπορούμε να αρχιοθετήσουμε με μεγάλο αριθμό πληροφοριών και δεδομένων, αλλά δεν, αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά δεν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ε, στη συνέχεια μια ερώτηση του κυρίου Μαχτά. Είπατε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Είπατε γιατί θέλουμε την καινοτομία και για ποιον θέλουμε την καινοτομία. Θέλουμε την καινοτομία διότι θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, θα έλεγα. Και θέλουμε την καινοτομία για όλους, είναι η απάντησή μου. Επιστήμη και καινοτομία για την κοινωνία, λοιπόν, για όλους για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες που δημιουργούνται από την παγκοσμιοποίηση. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα γίνει κατανοητό προς τους πολίτες. Είπατε ότι υπάρχουν τα πρωτότυπα, αλλά βρίσκονται ε, στα ε, γκαράζ, ε, βρίσκονται ε, κάπου σε ε, αφανή χώρο και με λυπεί αυτό το οποίο ε, είπατε και αυτό που συμβαίνει και είναι σημαντικό το ερώτημά σας όταν υπάρχουν οι καλές ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις όχι μόνο δημόσιες αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις και οι Υπουργοί έρευνα και Καινοτομία θα έπρεπε να είναι ταυτόχρονα και οι Υπουργοί Οικονομικών για να μπορέσουν να συνδυάσουν τι προσπάθειες ε, για τον τομέα που μα ενδιαφέρει. Προ την κυρία Νίμπλεχ τώρα, όσον αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, νομίζω ότι είμαστε πάνω από το στόχο. Είχαμε στόχο 20% και είμαστε στο 24% συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα. Τώρα, τι ποσοστό προέρχεται από τη βασική έρευνα, αυτό είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Συνήθως θέτω τέτοιου είδους ερωτήσεις στο ERC, γιατί αυτοί έχουν στατιστικά στοιχεία, πόσα έργα έχουν στο ERC, τα οποία μετασχηματίζονται σε αυτά έργα. Νομίζω ότι έχουμε 34 διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, από τον ε, έλεγχο ε, ιδεών που γίνεται στο ERC και νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια για το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο και για την καινοτομία για μια καλύτερη κοινωνία. και ξέρω ότι δεν έχω πλέον χρόνο, αλλά θα κλείσω μέσα σε δύο λεπτά. Θα επανέλθω με τα χαρά να συζητήσουμε για το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους τρεις πυλώνες αριστεία, ανοιχτό πνεύμα και αντίκτυπος. Προς τον κύριο Νίκα. Να σας τα πω και στα πορτογαλικά καλύτερα. επισκέφθηκα τις προάλλες ε, ε, μία επένδυση 1,3 δισεκατομμυρίων ε, για οχήματα υδρογόνου. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν έχουμε τις απαραίτητες επενδύσεις. Νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να δώσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις για να επιτύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω σύντομε απαντήσει προ τον Κλοντ Τούρμε για την ορατότητα των ενεργειακών πολιτικών. Για την ορατότητα των ενεργειακών πολιτικών, νομίζω ότι πρέπει αυτά τα οποία λέμε να τα κάνουμε πράξη. Δηλαδή, όταν μιλάμε ε, για την ενίσχυση της ενεργειακής στρατηγικής μας και λέμε ότι θα εξετάσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ε, ηλεκτρική κινητικότητα και το θέμα των μπαταριών, θα πρέπει η γλώσσα μας να είναι κατανοητή από τους πολίτες. Ο Μπερχάν Πικάχ μου είπε τις προάλλες γιατί δεν δημιουργείται μια ε, νέα ιδέα ότι ε, φτιάχνεται το πρώτο ηλεκτρικό αεροπλάνο παραδείγματος Χάιν. Ίσως βάζοντας ένα στόχο ο οποίος θα είναι κατανοητός και ορατός προς τα έξω μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο προς τους πολίτες. Ελπίζω να κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Ίσως μια ερώτηση από την κυρία Τόγια ε, δεν ε, απάντησα. Με άγγιξε η ερώτησή σας. Ξέρω ότι αυτά που είπατε δεν απευθύνονται μόνο σε μένα, αλλά πραγματικά ε, θέλω να έχω τις απόψεις σας για την έκθεση Καμπέσον Ουρής. Ελέγξτε το και δείτε ότι οι συστάσεις της έκθεσης θα μπουν σε αυτό αυτά τα οποία κάνει η Επιτροπή και θα είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε και να είμαστε υπόλογοι αν δεν ε, τα εντάξουμε στην πολιτική μας. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να τα λάβουμε υπόψη όλα αυτά. Και προς τον κύριο Γόιλ θέλω να πω ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας για το τι πρέπει να αλλάξουμε. Όταν τα πράγματα δουλεύουν σωστά, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που λειτουργούν σωστά και δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε. Στη βασική έρευνα κάνουμε πάρα πολύ καλά πράγματα που δεν πρέπει να τα αγγίξουμε, πρέπει να τα επαυξήσουμε αλλά όχι να τα αλλάξουμε. Αυτά που κάνουμε για θέματα εταιρικών σχέσεων και βιομηχανίας επίσης τα κάνουμε πάρα πολύ σωστά και δεν πρέπει να τα αγγίξουμε. Αλλά για κάποια είδη καινοτομία, αυτά που βλέπουμε ότι φεύγουν προς τις ΗΠΑ Πολιτείες ή άλλα μέρη του κόσμου, κάτι πρέπει να κάνουμε. Να συνενώσουμε λοιπόν όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας κάτω από ένα κοινό όνομα, ένα όνομα το οποίο θα αντικατοπτρίζει την καινοτομία στην Ευρώπη. Θα το λάβω υπόψη λοιπόν αυτό και όντως αυτά τα οποία λειτουργούν δεν θα τα αλλάξουμε. και προς την συμπατριώτησα μου, την, Μαρία, την κυρία Ματία, Μαρίζα Ματίας. Μπορούμε να τα πούμε και αργότερα, λέει η κυρία Ματίας. Όχι, ε, σίγουρα ε, το θέμα αυτό που είπατε και ο προβληματισμός σας για την επιστήμη τη συμπεριλήψη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μάλιστα πέρυσι Μία Κινέζα ε, προσωπικότητα ήταν το ε, βραβείο Νόμπελ ιατρικής που έλυσε το πρόβλημα της Ελληνοσία, ε, διαβάζοντας ένα ποίημα 2.000 χρόνων πριν. Οπότε υπάρχει σύνδεση της επιστήμης με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν θα πρέπει να την αγνοούμε. Και για την Άμυνα. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την άμυνα με το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 που είναι άσχετο με την άμυνα. Είναι σαφώ διαχωρισμένοι οι τομεί και σαφώ διαχωρισμένα κονδύλια. Κυρία, την κυρία Μούντι ξεχάσατε. Α, πολύ ωραία. Τελευταία φράση για την κυρία Μούντι και τον κύριο Κόχλιτσεκ. Για τα σιλό που είπατε, τις απομονωμένες έρευνες που γίνονται. Θα πρέπει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό και να έχουμε περισσότερη διατομιακή συνεργασία, περιλαμβάνοντας και τις κοινωνικές επιστήμες, να έχουμε ε, τους διδάκτορες ε, ιατρικής, ε, όσοι κάνουν διδακτορικό στην ιατρική, να λαμβάνουν υπόψη ή να παρακολουθούν και κάποια μαθήματα κοινωνικών επιστημών, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, να μην είναι απομονωμένοι οι κλάδοι και το κλίμα στα πανεπιστήμια μας θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα ολόκληρο. Επίσης είπατε θέλουμε καλύτερη επικοινωνία με τους Ευρωπαίους πολίτες. Και όταν απάντησα στον Κλωτούρμε για τι αποστολέ και τα νέα εγχειρήματα, αυτό εννοούσα. Καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη προβολή του έργου μα. Κύριε και ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Ελπίζω να μην άφησα πολλά έξω και να μην ξέχασα. Αλλά μπορούμε να βγούμε έξω και να σας απαντήσω κατηδίαν στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πολύ καλές απαντήσεις, αλλά τα κακά μαντάτα σας περιμένουν, γιατί ε, έχουμε στήσει την συνάδελφό σας, την κυρία Μπιενκόφσκα, που ξεροσταλιάζει 10 λεπτά μπροστά στην αίθουσα, περιμένοντας να τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Αγαπητοί φίλοι, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο Μπιενκόφσκα, που είναι αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, είναι εδώ στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Κυρία Μπιενκόφσκα, περιμένουμε την ενημέρωση και τα νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, στα θέματα αρμοδιοτήτων σας ε, του Προγράμματος Εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 και ε, τι μέλη γενέστε με το Πρόγραμμα Εργασιών του 2018. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε την πρότασή της για ένα πρόγραμμα για την βιομηχανική ανάπτυξη της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ξεκινήσει 2018 με 2020 με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε επίσης την διάμεση αξιολόγηση ε, σημαντικών προγραμμάτων όπως το Κόσμε, το Γαλιλαίο, το Κοπέρνικους. Περιμένουμε λοιπόν ενημέρωση και για αυτά τα θέματα και προοπτικές για το μέλλον αυτών των προγραμμάτων και ίσως και κάποιες πληροφορίες για τα μέτρα βιομηχανικής πολιτικής και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα μέτρα βιομηχανικής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά περιμένουμε με ανυπομονησία και σας δίνω το λόγο κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι ιδιαίτερως για την ευκαιρία που έχω να είμαι κοντά σας σήμερα. Δεν είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, αλλά ήταν το μόνο σημείο που είχα σήμερα, η μόνη υποχρέωση που είχα σήμερα, γιατί δεν είμαι και πολύ καλά. Θα ήθελα να πω κάποια γενικά λόγια για το τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα επικεντρωθώ σε τρεις ειδικού τομείς στους οποίους έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στους τελευταίους μήνες, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, ε, δηλαδή στο διάστημα, την άμυνα και την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρόσφατα ακούσαμε ε, ότι έχουμε ρωτά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει όμως να επαναπαυθούμε σε αυτές τις θετικές εξελίξεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δημόσιοι φορείς είναι να στηρίξουμε... Τι, τι, εγώ, εγώ, Uh, Θα πρέπει να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις και τους ε, Ευρωπαίους πολίτες με τις ε, πρωτοβουλίες μας. Μάλιστα, πρόσφατα ε, είχαμε το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση της παγκοσμιοποίησης, την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στη Χαλιβουργία και αλλού και επίσης θέλουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ε, το νέο, πανευρω... το νέο Πανευρωπαϊκό Ταμείο ε, του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου που περιμένουμε ως ούπο να λειτουργήσει. Ε, ασχολούμαστε και με τα θέματα των δεξιοτήτων μέσω του θεματολογίου νέων δεξιοτήτων. Και φυσικά προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την ε, λειτουργία της ενίας αγοράς μετά τη δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες, τη δέσμη μέτρων για τη συμμόρφωση και αμέσως μετά το καλοκαίρι ε, θα εγκρίνουμε και τη δέσμη μέτρων για τη συμμόρφωση στον τομέα των εμπορευμάτων και θα γυρίσουμε και την πρωτοβουλία μας για τις νεοφυείς και επεκτηνόμενες επιχειρήσεις. Αλλά έχουμε δράσει και σε επιμέρους τομείς και σε αυτό θα ήθελα να επικεντρωθώ και να σα ενημερώσω για τι τελευταίε εξελίξει στους τρει κλάδους που σα ανέφερα. Ξεκινούμε από το διάστημα. Τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίασα την ε, νέα μα στρατηγική για το διάστημα, που είναι περιεκτική και εμπεριστατωμένη και για πρώτη φορά έχουμε μια τέτοια ευρεία στρατηγική που ήδη αποφέρει καρπούς. Ε, καταρχήν τα προγράμματα Κοπέρνικος και Γαλιλαίος ήδη είναι λειτουργικά και τα χρησιμοποιεί η βιομηχανία και οι δημόσιες αρχές αλλά και ε, μεμονωμένοι πολίτες. Και του χρόνου θα επικεντρωθούμε στα θέματα ενίσχυσης της αγοράς, θα στηρίξουμε τις νεοφύσεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του διαστήματος, όλες οι νεοφύσεις είναι ούτως ή άλλως σημαντικές, θα προετοιμάσουμε την εξέλιξη του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου προς ε, νέες ε, προτεραιότητες, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, η ασφάλεια και άμυνα, Επίσης, ε, στα θέματα κλιματικών αλλαγών πρωτοστατούμε σε, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Θέλουμε να βελτιώσουμε την επιτήρηση και την παρακολούθηση του διαστήματος και να αξιολογήσουμε την ε, ε, πιθανή ε, νομοθετική πρωτοβουλία των κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών και να αναπτύξουμε μια έξυπνη στρατηγική για τους εκτοξευτήρες προκειμένου να έχουμε αυτόνομη πρόσβαση της Ευρώπης ε, στο διάστημα και γι' αυτό χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς εκτοξευτήρες και ενώ την Ariane 6 και το Vega C. Επίσης θα πρέπει να δράσουμε στα θέματα της διακυβέρνησης του τέστην θα πρέπει να δρούμε συλλογικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να μην χρονοτριβούμε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη της Επιτροπής σας προς τη στρατηγική μας που έχει πια αρχίσει να αναπτύσσεται και τα αποτελέσματά της ε, αρχίσουν να γίνονται όλο και περισσότερο ορατά από φέτος. Και φυσικά έχουμε και το σχέδιο της τελικής έκθεσης της κυρίας Κρέλ που μας βοηθά ιδιαιτέρως. Τους επόμενους μήνες θα χρειαστώ όλους σας την υποστήριξη για την εφαρμογή της στρατηγικής και φυσικά και στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι μεταξύ μας. Θα υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας μόνο εφόσον έχουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Θα σας ενημερώσουμε και για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος μας για το διάστημα φέτος το, το φθινόπωρο, κάτι που θα πυροδοτήσει και τη, τη θεσμική προετοιμασία για τις επόμενες προτάσεις. Παίρνω στους υπόλοιπους κλάδους ένα θέμα που με απασχολεί καθημερινά τους τελευταίους μήνες. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής, όπως θα έχετε διαπιστώσει, στο θέμα της ε, άμυνας. Πριν από δύο εβδομάδες ε, εγκρίναμε το πακέτο της άμυνας με τρία σημαντικά στοιχεία. Καταρχήν, έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Πρόκειται για ένα έγγραφο στρατηγικής προκειμένου να ε, ε, ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Συνεργασίας. Δεύτερο έγγραφο του πακέτου, η ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που ξεκίνησε πέρυσι. Και με την ανακοίνωση αυτή παρέχουμε πληροφορίες για το πεδίο εφαρμογής της προτεραιότητας και τη λειτουργία του Ταμείου αυτού για την άμυνα. Και τρίτο σημείο στο οποίο θα εστιαστώ σήμερα, ε, τον κανονισμό τμήμα του Ταμείου Άμυνας που θεσπίζει ένα πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ για μία διετία. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια της προοπτικής είναι το 2019 και 2020 του, των πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και μάλιστα την ίδια μέρα που έγινε λειτουργικό το Ταμείο Άμυνας είχαμε και τη δημοσίευση των πρώτων διαγωνισμών για τι προπαρασκευαστικές δράσει για την αμυντική έρευνα. Οπότε ε, έχουμε την ε, θέση εφαρμογή και του Ταμείου Άμυνας μετά την εκκίνηση της πρώτης φάσης των διαγωνισμών. Έτσι θα στρώσουμε το δρόμο για συγκεκριμένα ερευνητικά αμυντικά προγράμματα που θα προταθούν σε ένα χρόνο. Θα ήθελα επευκαιρία να σας ε, δώσω και κάποιες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Άμυνας, κάτι που είναι καινοτομία του πακέτου ένα πρωτοφανές ε, σημείο. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα για θέματα άμυνας. Κάτι ρηξικέλευθο και ανατρεπτικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα τη αμυντική μα βιομηχανία και γι' αυτό επιλέξαμε ω νομική βάση τη πρόταση αυτή το άρθρο 173 τη συνθήκη που αφορά την ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία. Και αυτό έχει κέρια σημασία γιατί αυτό που σκεφτόμαστε είναι αν θέλουμε ε, μακροπρόθεσμα να έχουμε μια αμυντική ένωση, χρειαζόμαστε μια στρατηγική αυτονομία στην Ευρώπη και για να την προωθήσουμε και για να την εξασφαλίσουμε χρειαζόμαστε μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανική αμυντική βάση, μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη και με το πρόγραμμα αυτό αυτό το στόχο εξυπηρετούμε. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του προγράμματο, θα καλύπτει ότι κυρίως στη φάση πρωτοτύπου, χθε το συζητήσαμε με κάποιους ε, εταίρους μας, ε, μάλλον είναι φάση ανάπτυξης καλύτερος όρος, ε, εκεί επικεντρώνονται οι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά την αλυσίδα αξία, στη φάση του σχεδιασμού της ανάπτυξης προσπαθούμε να μειώσουμε τους κινδύνους και να δώσουμε ενάψματα για τη συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, όπως σας είπα, αφορά το 2019 και 2020. Πριν πρόκειται για μια δοκιμαστική φάση, πριν υποβάλουμε ένα πιο περιεκτικό και περιστατωμένο πρόγραμμα για μετά το 2020. Σε ό,τι αφορά τα μέσα παρέμβαση, θα συγχρηματοδοτήσουμε με επιχορηγήσει το πολύ μέχρι 20% του συνολικού κόστου. Το υπόλοιπο ποσό θα εξασφαλιστεί από τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου και πιο δύσκολο είναι να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για την υποβολή των σχεδίων. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις από δύο τουλάχιστον κράτη-μέλη που θα υποβάλουν κοινά προγράμματα θα αποφύγουμε τις επικαλύψεις ε, με ισχύοντες θεσμικού φορείς και όργανα και η πρόθεσή μας είναι όπως και στην έρευνα να αξιοποιήσουμε τις ε, ισχύουσες δομές και κυρίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αλλά μην ξεχνάμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια συνοδεύονται και από υποχρεώσει. Οπότε θα πρέπει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και να κάνει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική ισορροπία, και αυτή είναι σημαντική για την επιτυχία του προγράμματο, βέβαια θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι αυτό το πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν στρέφεται ή δεν έχει στόχο μόνο τη μεγάλη βιομηχανία, τα μεγάλα κράτα-μέλη. Βέβαια δεν θα επιβάλλουμε γεωεπιστροφή, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε επιχειρήσει επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη-μέλη να μπορούν να υποφεληθούν από το πρόγραμμα. Και θα πρέπει η αμυντική βιομηχανία να ανοίξει την αλυσίδα εφοδιασμού στην διασυνοριακή συνεργασία, ώστε να έχουμε μια γνήσια ενιαία αγορά της άμυνας ε, στα, στα πλαίσια και του τρίτου πυλώνα του σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Γι' αυτό και ένα τμήμα του προπολογισμού θα το αφιερώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια αυτή η ισορροπία θα εξαρτηθεί και από τα σχέδια που θα συγχρηματοδοτήσουμε. Τέλος, για τα 500 εκατομμύρια ευρώ που προτείνουμε ως προπολογισμό, ξέρω ότι το θέμα αυτό έχει αρχίσει να γύρει πολλά ερωτηματικά. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το περιορισμένο περιθώριο λιγμών που έχουμε στο τρέχον πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, στον προπολογισμό μα, δηλαδή. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στην αμυντική μα συνεργασία, θα πρέπει να προβλέψουμε και επαρκεί πόρου για την συνεργασία αυτή. Και μάλιστα να το κάνουμε και γρήγορα. Με το πρόγραμμα αυτό, γιατί όπως ξέρετε δεν ασχολούμαστε με το πρόγραμμα αυτό παραπάνω από ένα χρόνο, αλλά περιμένουμε κάποια αποτελέσματα ήδη στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού. Και μάλιστα προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε φρέσκο χρήμα από τα περιθώρια και μία μεταφορά κονδυλίων από τις υπάρχουσες δημοσιονομικές γραμμές. Δεν θέλουμε όμως καθυστέρηση κανένα από τα τρέχοντα σχέδια, ούτε να διακυβευθεί η δρομολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων ή, ή τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον, θα προτείνουμε στην έρευνα αύξηση του προπολογισμού του προγράμματο. σημαντική αύξηση ενό δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως μέχρι το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται δηλαδή για μια πρωτοφανή και ταχύτατη κίνηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τώρα να εναπόκειται στου συνομοθέτε να παρακολουθήσουν αυτό το ταχύ ρυθμό και να επιδείξουν το ίδιο επίπεδο φιλοδοξία. Ελπίζω να μπορώ να υπολογίζω στη δική σα υποστήριξη, στην υποστήριξη τη Επιτροπή Ήτρε. Τώρα χρειαζόμαστε και άμεσες ταχείες διαπραγματεύσεις. Αν θέλουμε το πρόγραμμα να λειτουργήσει από τις αρχές του 2019, χρειαζόμαστε και πολιτική συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα και καλά σχέδια και προγράμματα από τα κράτη-μέλη ήδη από τις αρχές του επόμενου έτους. Γνωρίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά μια και έχουμε πάρει φόρα και δεν υπάρχει αντίσταση από κανένα κράτος μέλος και μια και η άμυνα πραγματικά μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστεύω τα Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της επίσπευσης του θέματος αυτού για να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα, απευθύνω αυτή την έκκληση και το κάνω καθημερινά προς τους υπουργούς εν ώψη και του, της Συνόδου Κορυφής της ε, εβδομάδας αυτής. Θα πρέπει να δράσουμε τάχιστα με συγκεκριμένα και φιλόδοξα προγράμματα που θα συγχρηματοδοτήσουμε. Επίσης, θα, ας μην ξεχνούμε ότι και οι προπαρασκευαστικές δράσεις της έρευνας και το πρόγραμμα ανάπτυξης είναι πιλωτικά σχέδια. Σήμερα δοκιμάζουμε την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στον κλάδο και έτσι θα προσδιορίσουμε στη συνέχεια πρώτα την διακυβέρνηση, μετά τις μεθόδους, μετά τους κανόνες, να δούμε αν είναι κατάλληλοι εν ώψη και του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα είναι η λίθος και για την ικανότητα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συζήτηση, διαπραγμάτευση και ελπίζουμε και συμφωνία για ένα τέτοιο θέμα που αφορά την άμυνα, συγγνώμη, ένα τέτοιο πρόγραμμα που αφορά την άμυνα. Οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια της αποτυχίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουμε. Τώρα για τον ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία. Το GR 2030 και η σχετική ομάδα υψηλού επίπεδου θα ολοκληρώσει το έργο της και τον Οκτώβριο θα υιοθετήσει την τελική έκθεση με συστάσεις πολιτικής. Οι συστάσεις αυτές δεν θα φορούν μόνο ε, την, τα αυτοματοποιημένα συνδεδεμένα οχήματα με μηδενικές εκπομπές. Θα εξετάσουμε και το θέμα των αυτόνομων αυτοκινήτων. Για αυτό το θέμα βέβαια έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας και ίσως η κοινωνία μας δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμη για τέτοιου είδους αυτόνομα αυτοκίνητα, αλλά κατά τη γνώμη μου, που ασχολούμαι, ασχολούμαι με το θέμα αυτό το τελευταίο χρόνο και, η αυτόνομη οδήγηση είναι πραγματικά βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής και θα έχει θεμελιώδη σημασία στο μέλλον. Γι' αυτό και θα υποβάλω συγκεκριμένες απτές προτάσεις για την περίοδο μέχρι το 2030. Ίσως είναι καλύτερο το κλίμα για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή για την ανάγκη ταχείας πρόοδου στην Ευρώπη. Σίγουρα όμως, γι' αυτό θα χρειαστούμε να ξεπεράσουμε πλήρω το σκάνδαλο με τις εκπομπές και με προβληματίζουν τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα που θα έχει τους καταναλωτές και την βιομηχανία. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα θα είναι ακόμη χειρότερα, γιατί πυροδότησε πολιτικές συζητήσεις για απαγορεύσεις των πετρελοκίνητων αυτοκινήτων. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε ταχύτατη κατάρρευση της αγοράς ε, δίζελ αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα στερήσει απλώς τη βιομηχανία από τα απαραίτητα κονδύλια, ε, ώστε να επενδύσει σε οχήματα μηδενικών εκπομπών. Και το έλεγα αυτό από την αρχή, συνεχίζω να το υποστηρίζω. Γι' αυτό Καλό τη βιομηχανία να λάβει συμπληρωματικά εθελοντικά μέτρα για τη μείωση των οξυδίων του αζότου, των εκπομπών οξυδίων του αζότου στο, στα υπάρχοντα διζελοκίνητα αυτοκίνητα και αν θέλει να σώσει την βιομηχανία του ντίζελ θα πρέπει η βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία να λάβει δράση και να αντίνει τις προσπάθειές της, γιατί μέχρι στιγμής δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα, αποτελέσματα. Τέλος, πολύ σημαντικό όμως θέμα, είχαμε ελπίζω να το νιώσετε κι εσείς έτσι, πολύ κακοφόρα συζήτηση την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και έχουμε μια συνεκτική κοινή στρατηγική για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτό άλλωστε ζητούσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τόγια για την ερώτηση που έθεσε και που έδωσε τη για τη συζήτηση. Ξέρετε, αλλά θα επαναλάβω ότι έχουμε πολλές στρατηγικές που επικεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή ε, Βιομηχανία. Ενία αγορά για τη στρατηγική, την, ψηφιακή αγορά, την ένωση κεφαλαίων, το πακέτο για την κυκλική οικονομία. Έχουμε περιλάβει τη βιομηχανία σε όλους τους κλάδους των πολιτικών μας και θα το επαναλάβω. Ε, και κατανοώ τις σας για την ανάγκη συνεκτικής στρατηγικής. Το είπα και ελπίζω καθαρά και εξάστερα και να το να έγινε αντιληπτό και στο Στρασβούργο, ότι είμαι υπέρ μια ενιαία ε, περιεκτική ε, και ευρεία στρατηγική για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ελπίζω να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μέχρι το τέλο τη θητεία μα. Γνωρίζω βέβαια από ενασχόληση με πολλέ στρατηγικέ ότι η οριζόντια συμπερίληψη της, βιομηχανικής, ε, της βιομηχανίας όλα τα έγγραφα είναι ένα, μια πρόταση που έχει οριμάσει γιατί έχουμε καλή γνώση, καλά στοιχεία και καλή συνεργασία με όλου του ενδιαφερομένου. Οπότε συντρέχουν οι προποθέσει για την οριζόντια συμπερίληψη τη βιομηχανία σε όλε τι πολιτικέ. Πάντω χρειάζομαι και τη δική σα βοήθεια και ε, υπολογίζω στην συνδρομή σας. Τώρα, να ολοκληρώσω. Τι μας απομένει για το υπόλοιπο μισό της Τα αποτελέσματα. Να δείξουμε έργο. Υπάρχουν στρατηγικές, οι δέσμες μέτρων, υπάρχουν και η στρατηγική για το διάστημα που φέρει καρπούς. Θέλουμε όμως απεγνωσμένα αποτελέσματα, ορατά αποτελέσματα. Δεν αρκεί, ούτε είναι σωστό να μιλούμε για την ανάγκη της ενιαίας αγοράς και μετά να αποδυναμώνουμε κάθε πρόταση που υποβάλλουμε. Δεν είναι σωστό να είμαστε υπέρ της αυστηρής εφαρμογής και μετά να προβάλλουμε αντίσταση όποτε θίγονται ένομα συμφέροντα. Ούτε είναι σωστό να μιλούμε για προώθηση της βιομηχανίας 4.0 και μετά να εισπράττουμε προστατευτισμό αντίστοιχο. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα μισή χρόνια που μας έχουν μείνει για να αποφέρουμε ορατά και καλά αποτελέσματα στις στρατηγικές και τις προσπάθειές μας. Και λυπάμαι που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας. και για τις πληροφορίες που μας δώσατε για το πρόγραμμα εργασιών για το τρέχον έτος. Να δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Κάριντς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Αν εξετάσουμε το παρελθόν των αμυντικών και στρατιωτικών κλάδων της βιομηχανίας, πολλές φορές ε, παίζουν πρωτοπόρο ρόλο στην έρευνα. Κάποιες τεχνολογίες από τις στρατιωτικές εφαρμογές περνάνε σε μη στρατιωτικές και έχουν ε, μεγάλη απόδοση αυτές οι επενδύσεις. Εγώ ως φοιτητής εργαζόμουν για τεχνολογίες ε, αναγνώρισης φωνής που χρηματοδοτούσαν ε, αμερικανικοί φορείς, τώρα λέγονται Siri και αρέσουν σε όλους. Αρχικά δεν χρηματοδοτείται αυτή η έρευνα από την Ευρώπη αλλά από τις ΗΠΑ. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι για να βοηθήσουμε την οικονομία μας, για να βοηθήσουμε τους διάφορους κλάδους να είναι ανταγωνιστικοί έναντι των ΗΠΑ πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα όχι μόνο στο διάστημα, στον κλάδο του διαστήματος αλλά και τον αμυντικό κλάδο. Πολύ σωστό αυτό. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Τώρα μια ερώτηση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι πολύ σημαντικός κλάδος και πολύ σημαντικό θέμα. Αναφερθήκατε στα αυτόνομα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς δηλαδή και αυτοκίνητα με μηδέν εκπομπές, μηδενικών εκπομπών. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Αλλά ξέρουμε ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία παράγει και πολύ οχήματα πολλά εσωτερικής καύσης και κυρίως κινητήρων δίζελ, όπου είμαστε πρωτοπορία. Εμείς αναπτύξαμε αυτούς ε, τους κινητήρες δίζελ με βάση και τους κλιματικούς στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Βέβαια έχουν υπάρξει διάφορες εταιρείε, ε, ξέσπασε το σκάνδαλο, μια σειρά από ό,τι φαίνεται, είτε κατάφορα ή σχεδόν κατάφορα παραβίασαν την ενωσιακή νομοθεσία. Αλλά Έχουμε τον έλεγχο και την έγκριση τύπου που ήταν ανεπαρκής σε επίπεδο κρατών μελών. Εφόσον εσείς είστε θεματοφύλακες και παρακολουθείτε πώς εφαρμόζονται οι κανονισμοί, τι θα αλλάξει σε επίπεδο Επιτροπής, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη συμμορφούνται με τις προδιαγραφές αυτές. Είμαι μέλος της πολύ ενδιαφέρουσα Επιτροπής για τις εκπομπές. Από ό,τι φαίνεται, ο ρόλος των κρατών μελών και ο ρόλος της Επιτροπής για να ελέγχουν αν εφαρμόζεται νομοθεσία είναι πολύ σημαντικός. Και των δύο. Για να διατηρηθεί, και αυτό είναι το σημαντικό, η εμπιστοσύνη του κοινού. Γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις ε, ατμομηχανές της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας και ένα τομέα όπου γίνονται πολλέ ε, καινοτομίε. Για παράδειγμα, αυτά τα αυτοκίνητα χωρί οδηγού και πολλέ άλλε καινοτομίε. Τι κάνουμε λοιπόν από πλευρά επιτήρηση για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων και άλλων καταναλωτών. Τόι από πλευρά των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Δεν θα μιλήσω για την άμυνα παρά το ότι είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα και έχει φυσικά και εφαρμογές ε, μη στρατιωτικές. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά δεν θα το θίξω. Θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Μαζί με τον κύριο Μπούτιχόφερ ε, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό και αυτό έχει επιπτώσει και στη χώρα μου και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι πέρασαν σε προγράμματα 4.0. γιατί όλα αυτά τα προγράμματα έχουν πολλές ε, εφαρμογές και σε άλλους τομείς, κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές εκ των οποίων δεν αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να κάνουν ένα τεράστιο βήμα, να περάσουν σε ψηφιακές μεθόδους εργασίας, να αλλάξουν τρόπους εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε τους αναγκαίους χώρους, για να ε, γίνει αυτή η συζήτηση ε, όπου αναφερόμεθα για παράδειγμα πως το κείμενο σε χώρους ψηφιοποίησης, σε κέντρα προώθησης ε, της καινοτομίας. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε αυτές οι ιδέες να προωθηθούν συντονισμένα. Οι μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του οικονομικού ιστού στην Ήπειρό μας πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνονται καλύτερα για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να τους δώσουμε συνεχή βοήθεια, συνεχή στήριξη. Και αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε μόνο στα κράτη-μέλη. Είμαι πεπισμένη ότι ακόμη και αν είχαμε 27 πολύ καλά εθνικά προγράμματα για το 4.0, δεν θα είχαμε σε κλίμακα ένωσης προστιθέμενη αξία. Πολλά μπορούμε να κερδίσουμε εντοπίζοντας και στηρίζοντας ε, τους τρόπους και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προωθήσουμε αυτές τις αλλαγές. Δεύτερον, πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο ρόλο του κέντρου. Πολλά από τα προγράμματά μας αναφέρονται σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Πρέπει όμως να δοθεί και άμεση και έμεση στήριξη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση και άλλα προγράμματα να βοηθούν την οικονομία. Βεβαίως η ψηφιοποίηση και η έρευνα και η γενοτομία βοηθούν την οικονομία. Καλούμε λοιπόν την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα γίνονται επαρκείς προσπάθειες για να ενθαρρύνουμε την έρευνα προς όφελος όλων και που θα επιτρέπει ε, να γίνει ε, ριζική μετατροπή ορισμένων κλάδων της οικονομίας μας. Πρέπει να το κάνουμε. Για να υπάρξει θετική αλλαγή χρειάζονται βοήθεια όλοι. Για παράδειγμα, ε, πρέπει να γίνει ενεργειακή αλλαγή και να υπάρξει και ποιοτική αλλαγή και για τα προϊόντα και για τις υπηρεσίες, γιατί υπάρχουν νέα περιθώρια για ε, την ε, νέα προσέγγιση για την οικονομία, που θα είναι λιγάκι περισσότερο παρεμβατική, δηλαδή κάτι που θα κάνουμε σε ένα κλάδο θα έχει επιπτώσει και σε πολλούς άλλους. Ούτω ώστε να βοηθάμε συνολικά την οικονομία, αλλά ιδιαίτερα την βιομηχανία. Χρειαζόμαστε μια νέα βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ για το ECR. Ο κύριος Τόσενοφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά είναι πάρα πολλές οι ασχολίες μα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω να καταφέρετε ε, όλα αυτά τα οποία μα παρουσιάσατε στο πρόγραμμα της διαστημικής στρατηγικής και ε, για τον Γαλιλαίο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα έργο όπου η Ευρώπη θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ηγετική θέση στην ε, τεχνολογία χρησιμοποιώντας ένα ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης. Ελπίζω να επιληθούν τα προβλήματα και για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού. Έχω και μία ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε για τις μεγάλες φιλοδοξίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχει μεγάλη πίεση ε, το συντομότερο δυνατόν ε, να αποκτήσουμε ε, αυτόνομα οχήματα, αυτοκινήτα χωρίς οδηγό. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μήπως τυχόν είναι πολύ γρήγορη αυτή η πορεία Ίσως θα, μπορέ, θα, θα ε, αφήνουμε τα ε, οχήματα ε, τα οποία ρηπαίνουν περισσότερο να βρίσκονται διαθέσιμα στην αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι όταν αναπτυχθούν τα νέα οχήματα. και να μας απασχολήσουν και άλλα θέματα όπως ε, η διάθεση των ε, ε, χρησιμοποιημένων μπαταριών και λοιπά όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Το ερώτημά μου είναι μήπως αν βιαστούμε υπερβολικά θα είναι πολύ δαπανηρή η νέα τεχνολογία για την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν θα είναι εφικτή και θα ήταν προτιμότερο ίσως να ακολουθήσουμε μια πιο αργή μετάβαση στη νέα τεχνολογία. Ίσως ε, μικρές ε, βιομηχανίες, ε, μικροί κατασκευαστές δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. Ο Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας και που μας παρουσιάσατε τις εργασίες της Επιτροπής και τα σχέδια της Επιτροπής. Μας ευχαριστήσατε διότι υποστηρίζουμε τη στρατηγική σας και σας διαβεβαιώνω ότι στην Επιτροπή μας ιδιαίτερα θα θέλουμε να σας υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο εάν έχετε και πιο ουσιαστική στρατηγική. Όσο περισσότερα έχετε να μας παρουσιάσετε, τόσο περισσότερο θα σας υποστηρίζουμε. Ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη όθηση από πολλούς τομείς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εστιαστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικότερα στην βιομηχανική πολιτική και έρευνα. Και αυτό διότι υπάρχει ο διεθνής ανταγωνισμός που αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε μας υποχρεώνει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ευρωπαϊκή έρευνα και βιομηχανία. Άκουσα την παρουσίασή σας και συμφωνώ με την ε, δήλωσή σας ότι θα χρειαστεί να έρθουμε αντιμέτωποι με δρεωμένα συμφέροντα κάθε είδους πρέπει να υπερασπίσουμε τη δική μας βιομηχανία έναντι κάποιων από αυτά τα δρεωμένα συμφέροντα που προβάλλονται ως υπερασπιστές της βιομηχανίας ενώ αντιθέτως οδηγούν την βιομηχανία μας σε αδιέξοδο. Υπάρχουν κάποια θέματα που πάντοτε ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας, όπως είναι το ενδιαφέρον μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να εξετάσουμε και το ρόλο που παίζει το ε, FDI, που παίζουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα βαδίζουν χέρι-χέρι και πρέπει η βιομηχανική πολιτική να συνδυάζεται με την εμπορική πολιτική και να μην αποτελεί απλώς προέκταση της εμπορικής πολιτικής. Και βέβαια πρέπει να εξετάσουμε και το δίκαιο του ανταγωνισμού. Όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, όπου καταβάλλεται μεγάλες προσπάθειες, θέλω να πω το εξή. Θεωρώ σημαντικό ε, να ε, προωθούμε την αμυντική βιομηχανία και υποστηρίζουμε αυτή την στάση, αλλά η προσέγγιση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά ε, θεραλέα, διότι ε, το να δίνετε 500 εκατομμύρια ε, κατέτος δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρήματα τα οποία θα εξοικονομούσαμε εάν είχαμε ισχυρότερους δεσμούς συνεργασίας. Η ίδια η Επιτροπή έδωσε αριθμητικά στοιχεία. Μας είπε ότι 25 με 100 εκατομμύρια το χρόνο θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν αν υπήρχε μεγαλύτερη συνεργασία. Και αυτό θα έπρεπε να τονίσουμε. Να, να εφαρμοστεί η οδηγία για τις συμβάσεις από το 2009 που θα μας έδινε μεγάλη όθηση και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι ακολουθείτε τις σωστές προτεραιότητες. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε αργότερα να το συζητήσουμε λεπτομερέστερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Συνάδελφος Κοχλίτσε από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, για, κυρία Επίτροπε, για την ε, εισαγωγική σας παρουσίαση που ήταν πληρέστατη. Όπως και στην συνάδελφος θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση για το πρόγραμμα Γαλιλαίο, γιατί το πρόγραμμα είναι σε λειτουργία, υπάρχουν ήδη δορυφόροι στο διάστημα και όλοι οι οργανισμοί που θα πρέπει ε, να ασχοληθούν με αυτό το θέμα έχουν σχετικά αιτήματα. Ε, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα είναι ενδιαφέρον για όλα τα κράτη-μέλη και θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι προθέσεις σας και τι μέτρα θα λάβετε για την προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς. πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε κι εμείς εξίσου ευέλικτοι όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί θα πρέπει πολύ γρήγορα να κινηθούμε. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική είναι μια επιτυχημένη στρατηγική και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ε, μιλήσαμε με την ε, Ένωση Βιομηχανών της Τσεχίας και ε, μας είπαν ότι ε, αυτό το πρόγραμμα θα αφορά μόνο τις μεγάλες χώρες και όχι τα μικρά κράτη-μέλη. Όλα ξεκινάνε από μια υψικάμινο. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται μια υψικάμινο και για τον τομέα του γυαλιού και για τον τομέα του χάλιβα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, θα υποστηρίξετε την καιροτομία και σε αυτόν τον τομέα που είναι κλειδί για όλες τις βιομηχανίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βαν Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είστε εδώ. Παρά το ότι ό,τι μας είπατε είστε λίγο αδιάθετοι. Να κάνω μερικές παρατηρήσεις ε, για το κλάδο βιομηχανίας, όπως τα περιμένατε. Γιατί όπως ακούσατε, είχαμε μια ειδική επιτροπή που έκανε, όπως είπατε, μια πολύ καλή έκθεση. Η ειδική επιτροπή μας, λοιπόν, που στηρίχθηκε από την ε, ευρία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η επιτροπή. Αλλά αυτά τα οποία εγκρίναμε δεν πρέπει να μείνουν στα χαρτιά. Όλοι οι συνάδελφοι δούλεψαν ε, πολύ σκληρά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερο είναι να εφαρμόζουμε αυτά που αποφασίζουμε ως Κοινοβούλιο. Είστε η πρώτη ε, ε, παραλήπτης των παρατηρήσεών μας. Είστε η Επίτροπος που ασχολείται με τα δικά μας θέματα για να εφαρμόσει αυτά που αποφασίζουμε. Τα πρώτα θέματα είναι για την για τον ε, παράγοντα συμμόρφωσης. για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι άργησε πάρα πολύ η εφαρμογή του Euro 6 παρά το ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το παράγοντα συμμόρφωση. Πρέπει αυτό να αλλάξει. Το παρόν έτος θα πρέπει να είναι το έτος αναθεώρησης, τροποποίησης αυτού του παράγοντα συμμόρφωσης. Οπότε πρώτη ερώτηση, τι γίνεται με αυτό κύριε Επίτροπε, υπάρχουν προτάσεις για να αλλάξει. Τα άλλα δύο θέματα είναι αλληλένδετα και συνδέονται και με αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας. Θα πρέπει να πω ότι μάλλον διαφωνώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες εθελούσιες προσπάθειες σε αυτό το τομέα. Όχι. Ο κλάδος δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει ούτε καν ε, ε, την ομοθεσία. Τώρα να περάσουμε σε εθελούσιες προδιαγραφές δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και περιέχεται και στην έκθεση της ειδική επιτροπή, είναι να εισαχθεί η νέα προδιαγραφή, το Euro 7. Και να σας δώσω ένα επιχείρημα υπέρ αυτής της άποψη Μέχρι το 2023 και οι Ηνωμένε Πολιτείε, αμάν, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα θα έχουν πιο φιλόδοξες ε, προδιαγραφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο λοιπόν από περιβαλλοντική άποψη και για την ποιότητα του αέρα, αλλά και προς το συμφέρον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Χρειάζεστε ισότιμο ανταγωνισμό όσο γίνεται. Θα έπρεπε λοιπόν να εισαχθεί η προδιαγραφή Euro 7. Άρα είναι πολύ σημαντικό κύριε Επίτροπε να υποβάλλετε νέα πρόταση γι' αυτό. Και θα στηριχθείτε από την ε, Ευρία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, αν λάβετε υπόψη την Επιτροπή μα και τα απορίσματά τη Τελευταία. Μηδενικέ εκπομπέ, τι αναφέρατε. Αλλά είπατε ότι εθελουσίω θα καταλήξουμε. Ελπίζουμε να υπάρχει ένα νέο ε, μια νέα νομοθεσία για το διοξιδίο του άνθρακα μέσα στο πακέτο κινητικότητα. Θα υπάρξει μια πρόταση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εθελούσια η προδιαγραφή. Θα πρέπει να είναι δεσμευτική σε αυτή την νομοθεσία ότι θα έχουμε οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως υπάρχει ήδη σήμερα στην Καλιφόρνια, για να πιέσουμε τον κλάδο προς τη σωστή κατεύθυνση. Να τους υποχρεώσουμε να περάσουμε πολύ περισσότερο στα ηλεκτρικά οχήματα. Θα το στηρίξετε. Ευχαριστώ, ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μία ερώτηση που θα μπορούσε να απαντηθεί με απλό τρόπο. Χθε νομίζω ή προχθέ η ΙΝΤΑ ψήφισε μια συμφωνία για μέτρα anti-dumping, πώς θα αντιμετωπίσουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Και νομίζω ήταν ε, καλά ισορροπημένη αυτή η πρόταση γιατί στηρίχθηκε από πολύ ευρία πλειοψηφία. Θα τη στηρίξετε την έκθεση αυτή. Γιατί όταν θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος όλοι αυτοί που λένε ότι πρέπει να στηρίξουμε πολύ τον κλάδο θα προσπαθήσουν να αποδυναμώσουν την ε, πρότασή μας. Οπότε η ερώτησή μου θα είστε στο πλευρό μας να στηρίξετε την έκθεση ίντα. Είχε γίνει και στην Επιτροπή μας εδώ ήτρε ένα τμήμα της εργασίας για να καταλήξει αυτή η έκθεση. Δεύτερο θέμα, κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα θα μας βοηθήσετε να πείσουμε την κυρία Βέσταγκερ να επανακαθορίσει ποια είναι η κατάλληλη αγορά. Γιατί βεβαίω την εκτιμώ, είναι ευφιέστατη. Όλη η Επιτροπή γνωρίζετε ότι σήμερα ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. Η Επιτροπή πάντα μοιάζει να εκπλήσεται όταν μια επιχείρηση κατέχει κυρίαρχη θέση, αλλά δεν βλέπουμε ότι η Κίνα κατέχει πάνω από 50% της αγοράς και δεν κάνουμε τίποτα. Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν νέοι βιογνωμικοί κλάδοι, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε τους υπάρχοντες. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η συνάδελφος Φαν Μπρέμπτ. Μηδενικές εκπομπές. Η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα θα, θα συνεχίσει να αυξάνεται με πολύ ψηλό ρυθμό. Δεν ξέρω αν θα είναι σε 5 ή 10 ή 15, αλλά όσο νωρίτερα το αντιμετωπίσουμε, τόσο καλύτερα. Νομίζετε ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος εκπομπών μας δίνει τα κατάλληλα μέσα για να ενθαρρύνουμε επενδύσεις, εγώ αμφιβάλλω και μάλιστα ιδιαίτερα. Και τελευταίο, που συνδέεται και με τη ζήτηση που κάναμε και με τον κύριο Μουέντας, τι θα κάνουμε για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βοηθάει πολύ η Ευρώπη την έρευνα και την τεχνολογία και δυστυχώς όπως βλέπετε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλού φτιάχνουν τις μπαταρίες. Πώς θα κάνουμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσω για την επαναβιομηχάνηση για να βοηθήσουμε την καινοτομία, για να γίνεται παραγωγή εκεί που δώσαμε τις πρώτες οθήσεις μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τούρμες είναι ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, για το Dieselgate, για το σκάνδαλο, ε, πραγματικά ε, ήταν πολύ ανώμαλη προσγείωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όταν ήρθατε στην Επιτροπή, Φαίνεται, κάνατε σαν να μην είχατε διαπιστώσει το μέγεθος, την έκταση της απάτης. Σήμερα φαίνεται ότι το συνειδητοποίησατε και η Γερμανία στο Αποφασιστικό Συμβούλιο ήταν μειοψηφία και αυτό είναι καλό. Τώρα καλούμαστε να κάνουμε δύο πράγματα. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαδραματίσετε ένα κεντρικό ρόλο στην επιτήρηση της αγοράς Εγώ για πολλά χρόνια παρακολουθούσα το GRC Vela Lab και έχω την αίσθηση ότι χάνουν την ικανότητά τους από στιγμή σε στιγμή. Ενώ εμείς κερδίζουμε έδαφος ό,τι αφορά την επιτήρηση της αγοράς. Μπορείτε όμως να με διαβεβαιώσετε ότι η κακή διαχείριση του Vela Lab τους τελευταίους μήνες ε, θα διορθωθεί χάρη σε συνομιλίες που θα έχετε με τον κύριο Ναύρατση, τον Επίτροπο Ναύρατση. Δεύτερο θέμα, μπαταρίες. 35 με 40% της οικονομικής αξίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου βρίσκεται στην μπαταρία. Σήμερα η Ασία κυριαρχεί και η Ρωσία. Και εμείς είμαστε ουραγοί. Για τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα πρέπει να καταρχήν ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Πάντως για τις μπαταρίες ε, και να συνεργαστούμε και με την Nokia, με το εργαστήριο της Nokia. Αλλιώς, αν δεν συνεργαστούμε και αν δεν ανασκουμποθούμε, θα μείνουμε πίσω. Χρειαζόμαστε και στην Ευρώπη παραγωγή μπαταριών. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ε, με χρήματα του Ομπάμα κατάφεραν οι Αμερικανοί να νικήσουν τους ε, Ασιάτες, γιατί να μην ε, μπορέσουμε και εμείς ε, να κυριαρχήσουμε δημιουργώντας ε, ισχυρά εργοστάσια για να παρασκευάζουμε τις δικές μας μπαταρίες. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Παρακαλώ κυρίε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με το πακέτο της άμυνας. Ε, τη διτή χρήση. Για την έρευνα και για θέματα αμυντικά και για θέματα μη στρατιωτικά σίγουρα από πολλέ απόψεις η άμυνα πυροδότησε την καινοτομία στο Ιντερνετ για παράδειγμα, από εκεί προέκυψε. Και εμείς με το Ταμείο μας θέλουμε να κλείσουμε το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων περιοχών. Και θέλουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο και ε, επενδύοντας σε τέτοιες τεχνολογίες και ικανότητε στην άμυνα, σίγουρα θα καταφέρουμε να επηρεάσουμε θετικά και το μη στρατιωτικό κλάδο. Οπότε επικεντρωνόμαστε και στο σκέλος της έρευνας και στο σκέλος των ικανοτήτων. Γι' αυτό θέλω ε, να επισπεύσουμε τις εργασίες συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το τελευταίο εξάμεινο με μεγάλη επιτάχυνση. Και ακριβώς λόγω της, ε, των ξεχωριστών ε, συμβάσεων έχουμε ένα κενό 25 με 100 δις ε, το χρόνο. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα εξοικονομήσουμε με καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών στις προμήθειες. Έχουμε τώρα δύο ε, οδηγίες για τις προμήθειες στην άμυνα και τις μεταφορές. δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη ε, διαδικασίες έχουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα μόνο και συνεχίζουμε το διάλογο με τα κράτη-μέλη, γιατί γνωρίζουμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή από αυτή την άποψη. Αλλά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι το έργο μας σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης είναι άχρηστο. Γιατί θέλουμε να δώσουμε ενάψματα για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και όπως είπα πριν, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα τουλάχιστον και φαίνεται και από την εφαρμογή των δύο οδηγιών, το πιο δύσκολο θα είναι οι κοινέ ε, αγορέ, κοινέ προμήθειε. Και αυτό είναι προπόθεση για να λάβει κανεί το 20% τη χρηματοδότηση. Τουλάχιστον τρει επιχειρήσει από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη σε κοινά προγράμματα. Και φυσικά όσο περισσότερα κράτη και επιχειρήσει συμμετέχουν τόσο το καλύτερο. Έχουμε 500 εκατομμύρια, όχι ετησίω, 500 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Για τα δύο τελευταία χρόνια των του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Θέλουμε να δώσουμε ενάυσματα λοιπόν με αυτές τις προτάσεις. Και τις προάλλες ε, συζητούσαμε εκπροσώπους των Υπουργείων Άμυνα, που προσπαθούν να ετοιμαστούν για να συμμετέχουν. Η βιομηχανία είναι ήδη έτοιμη και οι κοινέ αγορές, οι κοινέ προμήθειες σε θέματα αμυντικά ε, θα ενθαρρυνθούν χάρη στο πρόγραμμά μας. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο και τη διασύνδεση διαστήματος και άμυνας ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την παρουσία τους στον αμυντικό τομέα. Μέχρι στιγμής το Γαλιλαίο ήταν και θα είναι στο μέλλον όλο και πιο ακριβές πρόγραμμα. Είναι το ακριβέστερο ε, και πιο τεχνολογικά προηγμένο ε, πρόγραμμα δορυφορικής ε, ε, πλοήγηση στον κόσμο. Και σίγουρα η παριθμόν ένα προτεραιότητα είναι η προώθηση του Γαλιλαίου στην αγορά. Και θα καταφέρουμε χάρη στο Γαλιλαίο να προωθήσουμε και την καινοτομία. Γιατί ήδη οι επιχειρήσεις παντού στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παράγει το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Οπότε το μείζον οικονομικό φέλος από το Γαλιλαίο ήταν και θα είναι ο τομέα downstream σε ό,τι αφορά τη σύνδεση ε, διαστήματος και άμυνας, ε, είπατε ότι οι τσιχικές εταιρείες θεωρούν ότι η άμυνα θα επικρατήσει σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτού του εργαλείου, αυτού του προγράμματος, αλλά νομίζω ότι είναι σαφής ε, οι διασυνδέσεις των δύο κλάδων άμυνας και διαστήματος. Ακόμη και χθες ζήτησα από τα κράτη-μέλη μεγαλύτερη συμμετοχή και από τη βιομηχανία το ίδιο μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί δεν θέλουμε να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να υποβάλουν σχέδια. Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν τι σχέδια θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Βιομηχανική Ανάπτυξη της Άμυνας. Αλλά κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες υπάρχουν. Και ακόμη και χθε προσπαθούσα να κινητοποιήσω το ενδιαφέρον των κρατών μελών επισημένοντας τη σχέση διαστήματος και άμυνας. Και σίγουρα έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση. Έχουμε και τα προγράμματα κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών, θα το ενισχύσουμε και αυτό. Δεν έχουμε ακόμη σχέδια. Αλλά πραγματικά δεν βλέπω κανένα κίνδυνο για τον τομέα του διαστήματος και την παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του διαστήματος. Όπως σας είπα, θα αφιερώσουμε ένα τμήμα του προϋπολογισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι μικρότερες επιχειρήσεις σε μικρότερες χώρες είναι σημαντικό αυτό το θέμα και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για σχέδια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και μικρότερες επιχειρήσεις και μικρότερες χώρες θα υποφεληθούν και από τη στρατηγική μας για το διάστημα και από το σχέδιο δράσης για την άμυνα και τη διασύνδεση και τη συνέργεια μεταξύ των δύο. Σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, ερώτηση Τόγια. Πρώτα θα πρέπει να εφαρμόσουμε το έγγραφο για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Δεύτερον, θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις εθνικές στρατηγικές ψηφιοποίησεις. Και για αυτούς τους λόγους θέλουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής θέλουμε προτυποποίηση που είναι πολύ σημαντική, ε, τεχνικές, ε, τεχνολογίες βασικής εφαρμογής, γενικής εφαρμογής, συγγνώμη, το είπα και στο Στρασβούργο, Θέλουμε ευθυγραμμισμένες κρατικές πολιτικές για διάφορους τομείς και μια συνεκτική βιομηχανική στρατηγική χρειάζεται και για την ψηφιοποίησή της και για να έχουμε επιτυχία σε πολλούς τομείς στην Ευρώπη. Και ένα τμήμα αφορά την οικονομία των δεδομένων. Θα πρέπει και οι νεοφύσμες επιχειρήσει επιχειρήσεις να πρωτοστατήσουν στην οικονομία των δεδομένων. Και αυτό το θέμα συνδέεται με το διάστημα, γιατί το πρόγραμμα Κοπέρνικος είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ε, μαζικών δεδομένων. Και θέλουμε μέσω αυτού του προγράμματος να δώσουμε πρόσβαση και στις νεοφύσεις επιχειρήσεις σε αυτά τα δεδομένα και μάλιστα και δωρεάν, δωρεάν δεδομένα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και μάλιστα με απλό τρόπο θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση. Περνάω τώρα στα αυτοκίνητα. Τι γίνεται με την έγκριση τύπου μετά την Επιτροπή εμείς. Φυσικά θα συνεχίσουμε και εγώ θα συνεχίσω την πολιτική εφαρμογής. Θα είδατε την επιστολή που έστειλα στη Volkswagen χθες. Εφαρμογή της πολιτικής, το ανέφερα και στην επιστολή. Η πρόταση για την έγκριση τύπου θα ξεκινήσει στη διαδικασία των τριμερών διαλόγων. Είχαμε κάποια καθυστέρηση, αλλά θέλαμε ήδη από αυτή την εβδομάδα να ξεκινήσουμε. Όπως είπα και στο παρελθόν, θέλουμε μεγαλύτερη εποπτεία ευρωπαϊκή. Χρειάζεται οπωσδήποτε καλύτερη ευρωπαϊκή και περισσότερη ευρωπαϊκή εποπτεία. Αλλά δεν θέλουμε να σφετεριστούμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών εδώ. Είμαι ξεκάθαρη. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Είχαμε την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου Gear 2030 ε, και μετά θα προτείνουμε ένα γενικό περιεκτικό πακέτο με πρωτοβουλία μας για τις μπαταρίες και την πρωτοβουλία μας για τις υποδομές για τη φόρτιση των μπαταριών. Γιατί τα οχήματα μηδενικών εκπομπών θα γίνουν πιο φθηνά να αυξήσουμε την παραγωγή. Αυτό κάνει η Κίνα. Είχε μαζική αύξηση της παραγωγής πέρυσι και φέτος. Επίσης έτσι θα κρατήσουμε ζωντανή και ανταγωνιστική την αυτοκινητοβιομηχανία μας. Γι' αυτό μετά την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου Gear 2030 θα προτείνουμε δύο πρωτοβουλίες. Παράγοντας τη συμμόρφωση. Κυρία Βαμπρέμπτ, συνεχίζουν οι τεχνικές ε, εργασίες στο θέμα αυτό και όπως υποσχέθηκα μέχρι το τέλος του έτους θα υποβάλουμε τα τεχνικά στοιχεία. Εθελοντικά μέτρα. Το είπα στην αρχή. Οικιοθελή μέτρα από τη βιομηχανία. Αν η βιομηχανία ή δεν κάνει καμία κίνηση ή κινηθεί με πολύ αργούς ρυθμούς όπως τώρα, θα αναλάβουμε και άλλες δράσεις συμπληρωματικές. Αλλά με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν μπορούμε να σημειώσουμε ταχεία πρόοδο. Έχουμε μόνο τη διαδικασία επιβολή κυρώσεων ή επιπαραβάση και αυτή είναι χρονοβόρα. Σε ό,τι αφορά το στόχο μηδενικών εκπομπών, εγώ είμαι υπέρ δεσμευτικών στόχων μηδενικών εκπομπών για τα αυτοκίνητα και για την Ευρώπη. Για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, για το GRC πρώτα, το κοινό κέντρο ερευνών. Το συζητάμε με τον Επίτροπο Ναύρατζιτς και με το έχετε επισημάνει επανειλημμένος. Ελπίζω να μπορέσω όσον να σας καθησυχάσω ότι θα εξομαλυθεί σύντομα η κατάσταση. Αυτό είναι ένα κενό που έχουμε στις εργασίες μας. Δεν, μπορώ να σας δώσω τώρα συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά ελπίζω ότι στο πολύ έγκυς μέλλον θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το GRC. Έχουμε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για τις μπαταρίες, όπως σας είπα και πριν. Και θα συνδέσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες με την Γερμανία, Ελβετία και Γερμανία με σεβασμό των εξαιρέσεων για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, συνεργαζόμαστε με τη Σισίλια Μάλστρομ για πιθανά μέσα ελέγχου των άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς, θα πρέπει να προστατεύσουμε την βιομηχανία μας και ταυτόχρονα να μην γυρίσει μπούμεραγκ αυτή η πρόταση. Τα κράτη-μέλη ήδη έχουν κάποια μέσα που τους επιτρέπουν να σταματήσουν ανεπιθύμητε ξένες αλλοδαπές αλλοδαπέ άμεσες αλλά πολλές φορές δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Και τα μέσα υπεράσπιση του εμπορίου, προστασία του εμπορίου συζητήθηκαν εκτενώς και στη Χαλιβουργία. Και ξέρετε πόσο χρονοβόρα είναι η συζήτηση στο Συμβούλιο των μέτρων προστασίας του εμπόριου που ήταν τόσο σημαντικά για τη χαλιβουργία μας. Και παρόλα αυτά η συζήτηση τράβηξε επί μακρόν. Κάποιες Άμεσε ξένε επενδύσει φυσικά είναι ευπρόσδεκτε σε μερικά κράτη-μέλη. Εμά δεν μας αρέσουν πάντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αντιβαίνουν στου στόχου τη ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι δύο όψει του ίδιου νομίσματο ουσιαστικά. Αλλά συνεργάζομαι στενότατα με την Επιτροπή Μάλστρομ για να ρυθμίσουμε το θέμα. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Με τόσα χαρτιά που είχα. Σας ευχαριστώ. Ε, Κυρία Επίτροπε, εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για τις δηλώσεις σας, για τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις. και είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα δούμε πρόοδο και στις δικές σας αρμοδιότητες, στην εσωτερική αγορά, την επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη διαστημική πολιτική. Όλοι είναι σημαντικοί τομείς για την πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νιώθουμε και εμείς υπεύθυνοι ε, γι' αυτό, όπως και εσείς είστε υπεύθυνοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους τομείς αυτούς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο στις 9 το πρωί θα έχουμε τον Επίτροπο Αρίας Κανιέτε. Οπότε θα είναι ε, καταπληκτική αυτή η αλληλουχία των Επιτρόπων Μοέντας, Μπιενκόφσκα, Κανιέτε. Οπότε ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 για τη συνέχιση με έναν καινούριο επίτροπο. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε.